Hello, good afternoon. Good afternoon, everybody. Καλησπέρα. Είχαμε προβλήματα οργανωτικά. que nadie de aquí ha ido y que desprecian, una cosa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 la actividad parlamentaria del IBE. Venga. Buen après-midi a todos. Buen après-midi. Καλησπέρα σε όλους. So, so, again, good afternoon. Για τρίτη φορά καλησπέρα. είστε εδώ, να σας δώσω μια εξήγηση. Η σύνοδος της ε, Επιτροπής ε, Ελευθεριών, η σημερινή, και η αυριανή ολόκληρη συνεδρίαση, κατά τύχη ε, συμπίπτει με μια πρωτοβουλία τριών Ευρωβουλευτήνων από την Επιτροπή Γυναικών. Υπάρχει μια χρονική σύμπτωση εδώ που κάνουμε αυτή την κοινή σύνοδο με την Επιτροπή Γυναικών και τη σημερινή που την κάνουμε μόνοι μας ως Επιτροπή Ελευθεριών. Δεν θέλω να ξανασυμβεί. Δεν είναι σωστός τρόπος εργασίας αυτός. έχουμε αυτό το πακέτο θυμάτων, ουσιαστικό θέμα και το διαπραγματευόμαστε μόνοι μας, ε, ενώ την ίδια στιγμή παράλληλα η Επιτροπή Γυναικών ε, ασχολείται πάλι με το ίδιο θέμα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά των θυμάτων να παραστούν εδώ. Είναι ατυχές αυτό. Φυσικά η εξήγηση είναι ότι για πρακτικούς και οργανωτικούς λόγους χρειάστηκε να οργανώσουμε έτσι τις ε, συνεδριάσεις μας. Δεν συνηθίζεται αυτό. Ζητώ την κατανόησή σας. Σας ε, διαβεβαιώνω ότι θα ξανασυμβεί. Προσπαθούμε να οργανώνουμε τις εργασίες μας με τρόπο σωστό. Δεν θέλουμε τέτοια πράγματα να ξανασυμβούν αυτές οι συμπτώσεις. Ελπίζω να σας ικανοποιεί ως εξήγηση. Πάμε στο σημείο 1, μετά από την εξήγηση, που είναι το σύνηθε σημείο έγκριση ημερήσιας διάταξης. Να σας πω ότι στο σημείο 7, για τις επιθέσεις κάτω των συστημάτων πληροφορικής, με εισηγήτρια την κυρία Χολμάιερ, αναβάλλεται το 17 η σύμβαση του Δουβλίνου θα το διεκπαιρεώσουμε στα πλαίσια του σημείου 2, στα πλαίσια των ανακοινώσεων του Προέδρου, το σημείο 18 για την ε, οδηγία για τις ε, συνθήκες ε, υποδοχής. Θα το διεκπαιρεώσουμε μαζί με τις ανακοινώσεις του Προέδρου και όχι σε χωριστό σημείο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν έχετε αντιρρήσεις, μπορούμε να συνεχίσουμε. Κύριε Μπουσουτήλ, κύριε Πρόεδρε προσυπογράφω αυτά που είπατε σε ό,τι αφορά τη σύμπτωση αυτών των συνεδριάσεων. Αυτή τη στιγμή γίνονται δύο διαφορετικές συνεδριάσεις Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ταυτόχρονα. Το οποίο είναι απαράδεκτο και σχιζοφρενικό. Δεν μπορούμε να είμαστε σε δύο διαφορετικούς τόπους παράλληλα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Υποστηρίζω αυτά που είπατε. Δεύτερον, είπατε ότι το σημείο 7 αναβάλλεται Θα ήθελα να συνεδριάσω τους συντονιστέ τότε, εφόσον ε, το σημείο αυτά δεν θα το διεκπαιρεώσουμε, 15 θα νωρίτερα. Του έχουμε πει να είναι εδώ σε 6.30. Α έρθουν ε, λοιπόν στι 6 και 4 για να τελειώσουμε και 15 λεπτά νωρίτερα. Η Ρενάτα Βέμπερ. Τη βλέπω μπορείτε να, ε, να στείλετε ένα μήνυμα και στους υπόλοιπους συντονιστές. Φαντάζομαι ότι και αυτοί θα θέλουν να τελειώσουμε 15 λεπτά νωρίτερα, εφόσον όμως αρχίσουμε 15 λεπτά νωρίτερα. Εντάξει, ας το έχουμε υπόψη μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε στη σημερινή συνεδρίαση, ούτως ώστε να προχωρήσουμε γρήγορα, να αξιοποιήσουμε σωστά το χρόνο μας, ούτως ώστε να τους συντονιστές τουλάχιστον για μία ώρα προβλέψαμε 45 λεπτά. Μπορούμε κάλλιστα να συνεδριάσουμε για μία ώρα. Μετά την απογευματινή συνεδρίαση συνεδριάζουν οι συντονιστέ λοιπόν. Όλοι μα λοιπόν έχουμε υπόψη μα τη συνεδρίαση αυτή των συντονιστών. Επίση να μην τελειώσουμε στι 6.30 την ε, τακτική μα συνεδρίαση, αλλά στι 6 και 4. 15 λεπτά νωρίτερα. Επαναλαμβάνω, τέτοιου τύπου πράγματα δεν πρέπει να συμβαίνουν συνήθω. Αλλά με το φόρτο εργασία, μερικές φορές είμαστε αναγκασμένοι να έχουμε ολομέλειες στο Στρασβούργο παράλληλα με τις συνεδριάσεις ε, της Επιτροπής μας. Όσοι λοιπόν ασχολούνται με την ολομέλεια δυσκολεύονται να παραστούν και στις συνεδρίες της Επιτροπής Ελευθεριών. The, Να συμμετάσχουν λοιπόν στις συζητήσεις και των δύο φόρουμ ταυτόχρονα. Θα προσπαθούμε να διορθώσουμε την κατάσταση, τόσο ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Πάμε στις ανακοινώσεις. Σημείο 2. Έχουμε τις διαπραγματεύσεις για την διαδικασία, για τις διαδικασίες, οι διατυπώσεις. Το Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση για την διαδικασία αυτή, ε, για την οδηγία αυτή στην 1η Απριλίου, 1η ε, Ιουλίου 2011 η Κομισιόν παρουσίασε την τροποποιημένη πρόταση που λαμβάνει υπόψη κάποιες από τις τροποποίησεις που είχε προτείνει το Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση και λαμβάνει υπόψη κάποιες από τις ανησυχίες του Συμβουλίου η πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, όπως υιοθετήθηκε στην Ολομέλεια του Απριλίου του 2011, ε, μας έδωσε και την διαπραγματευτική εντολή για την πραγμάτευση με το Συμβούλιο. Μετά όμως από την πρόταση την τροποποιηθήσα, η Σιλβίκη Γιώμ, η συγγήτρια και οι σκιώδεις συγγητές ε, είχαν διάφορες συνεδριάσεις για να υπάρξει μια νέα προσέγγιση για τα νέα τμήματα τη τροποποιηθή σα πρόταση τη Κομισιόν. Η άποψη των εισηγητών και σχεδόν εισηγητών μοιράστηκαν σε όλα τα μέλη τη ΛΥΜΠΕ. Θέλω να μου δώσετε την άδειά σα να στείλουμε ένα, μια επιστολή στη Δανέζικη Προεδρία και να παραπέμπουμε στη θέση τη πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου και στην άποψη στην οποία έχουν καταλήξει η Σλιβίκη Γιώμ και οι σκιώδης συζητητές για τα νέα τμήματα, εν ώψη των επόμενων διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Εάν δεν έχετε αντίρρηση σε αυτή την πρόταση, τότε θα στείλω επιστολή στη Δανέζικη Προεδρία, ΣΥΒΗ. Ευχαριστώ πολύ σύντομα. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο για αυτή την ανακοίνωση. Ευχαριστώ και τους κοιόδης εισηγητές που έδειξαν πνεύμα συνεργασίας και επιμονής αυτούς τους τελευταίους μήνες και εργατικότητας. Ευχαριστώ όλους όσους συνεργάστηκαν ε, στο εσωτερικό της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ, το προσωπικό της Επιτροπής μας και τους βοηθούς. Όπως είπατε Πρόεδρε, ε, δεν ήταν εύκολη ιστορία αυτή, αυτού του ντοσιέ και θα εξακολουθούμε να δυσκολευόμαστε εξαιτία του στο μέλλον. Λάβαμε τον Ιούνιο του 2011 για να βγούμε από το διέξοδο των διαπραγματεύσεων μια πρόταση νέα από την Κομισιόν, τροποποιηθήσα και το κείμενο αυτό επέφερε πάρα πολλέ ε, τροπολογίε από το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2011. Αυτό είναι και, αυτή είναι και η εντολή διαπραγμάτευσή μα με το Συμβούλιο. Υπήρχαν και τμήματα όμω επί της πρότασης της ε, Κομισιόν, όπου εμεί δεν είχαμε λάβει θέση ω Κοινοβούλιο. Ε, στα πλαίσια αυτή της κοινή προσέγγισης, λοιπόν, όμω το κάναμε. Για τα επόμενα στάδια τώρα, η Δανέζικη Προεδρία με ενημέρωσε ότι το Συμβούλιο δεν έχει εντολή και οι τεχνικές συνεδριάσεις ε, είχαν ε, καταλήξει. Οι πολιτικές συνεδριάσεις δεν έχουν γίνει όμως και δεν ξέρουμε αν ο πρώτος τριμερής διάλογο μπορεί να γίνει επί Δανέζικη προεδρία. Τέλο Δεν είναι μυστικό ότι πολλά κράτη-μέλη είναι αρνητικά. Έτσι, για να μην το πω και πιο έντονα, πιο ομά, για κάποια σημεία, για κάποιες πρόοδους. Εμείς ε, είμαστε στεναροί στο Κοινοβούλιο όμως, για το τι άλλαξε και για το τι μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Δεν θέλω να κάνω καμία παρήθμιση, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι δίνουμε μεγάλη σημασία, ιδίω στις ε, εγγύησει για τους μη συνοδευμένους ε, ανήλικους, για την εξέταση ποιότητας σε πρώτο επίπεδο, πρώτο πρωτοβάθμος, ε, για τους λόγους επιτάχυσης της ε, διεκπεραίωσης της ε, αίτησης, για την έννοια της ασφαλούς χώρας. Όλα αυτά τα συζητήσαμε πάρα πολύ και νομίζω ότι θα παραμείνω στη μέση διάταξη. Ευχαριστώ για αυτή την ενημέρωση που μας κάνατε. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος Σιλβή. Σας ευχαριστώ για τη θέση του Κοινοβουλίου όπως μας την παρουσιάσατε. δεδομένης της θέσης του Κοινοβουλίου προβλέπεται ότι θα υπάρξει εντολή Δανέζικης προεδρίας για μια διαπραγμάτευση για την πρώτη ανάγνωση του Συμβουλίου. Η πρόταση λοιπόν να γράψω στη Δανέζικη Προεδρία για να τις αναφέρω την θέση του Κοινοβουλίου. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό εγκρίνεται από την Επιτροπή μας. Πάμε στο επόμενο σημείο που είναι ο κανονισμό Δουβλίνο 2. Υπάρχουν κάποιε ε, πληροφορίες εδώ. Κυρία Φίξτρομ, μπορείτε να μας πείτε σύντομα ποια είναι η κατάσταση. Και μετά θα ακούσουμε από τον κύριο Αντώνιο Μασίπ, ο οποίος πρέπει να πάει στη συνεδρίαση της Νομικής ε, Επιτροπής. Κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας ενημερώσω σύντομα. η κατάσταση του φακέλου του πλήνω 2. Είχαμε δύο τριμερεί διαλόγους και υπάρχουν δύο ακόμα συνεδριά τριμερού διαλόγου για τον Ιούνιο. Η Δανέζικη Προεδρία ε, θέλει να καταλήξει συμπέρασμα πριν από το τέλος του Ιουνίου και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με τη Δανέζικη Προεδρία για να φτάσουμε στον τον πιο μακριά μπορούμε. Όμω το Κοινοβούλιο είναι αποφασισμένο να μην, διασυστεί, να μην για συμφωνία. Περιμένουμε τρία χρόνια το Συμβούλιο να έρθει και να μα πει τι αποφασίζει για το φάκελο αυτό. Α περιμένουμε λίγε εβδομάδε ή μήνε, αν χρειάζεται λοιπόν. Ούτω ώστε η συμφωνία που θα καταλήξουμε να είναι καλή. Περιμένουμε όχι μόνο μία συμφωνία, αλλά μια καλή συμφωνία υπάρχει πάντως καλή συνεργασία και πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τη Δανέζικη Προεδρία. Ευχαριστώ και την Προεδρία και όλους τους σκιώδους εισηγητές και το προσωπικό της ε, Επιτροπής, τους υπαλλήλους, για την καλή συνεργασία. Γι' αυτό προχωρούμε ομαλά, γρήγορα, προς μία καλή συμφωνία στο τέλος του τούνελ. Κάποια θέματα έχουν επιληθεί, αλλά θα ήθελα να σας πω για όσους ενδιαφέρεστε ότι το άρθρο 26 για τα ένδικα μέσα και το άρθρο 27 για την κράτηση ήταν τα πιο περίπλοκα θέματα και πρέπει να επιληθούν. Δεν έχουν ακόμα επιληθεί, είναι προς επίλυση. Το άρθρο 11 επίσης. Ή όπως λέει η θέση του Συμβουλίου, το άρθρο 16α για τα εξαρτώμενα μέλη, προβληματικά. Μια το, Μια και το Συμβούλιο τα έβασε επέβαλε στο τέλος της ιεράρχησης των κριτηρίων. Η κράτηση είναι οριζόντιο θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε περαιτέρω στους τριμερείς διαλόγους για, για την οδηγία των όρων υποδοχής. Για τα ένδικα μέσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ στεναρό. Όχι, δεν πρέπει να υπάρξουν μεταφορές πριν πριν ληφθεί απόφαση ε, για τον ανασταλτικό χαρακτήρα. Ευτυχώς το άρθρο 31 για το μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης είναι σχεδόν, έχει σχεδόν συμφωνηθεί και θα μας δώσει ένα νέο αποτελεσματικό εργαλείο για να παρακολουθήσουμε τα σύστηματα ασύλου στα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να αποφύγουμε ε, κάποιος κρίκος της αληθίδας να σπάσει. Ευχαριστώ ξανά όλους όσοι έχουν εμπλακεί σε αυτή την πολύ δύσκολη ιστορία, σε αυτό το δύσκολο φάκελο. Παραμένω στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, εφόσον έχετε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Κύριος Μασίπ, ο, οδηγία για τους όρους υποδοχής. Τι διεμήθη στον τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ. Είχαμε τη δεύτερη συνεδρίαση του τριμερούς διαλόγου. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και άλλη μια συνάντηση και κατά πάσα πιθανότητα και άλλη μια στις 19 του μήνα. Δεν είναι τόσο μεγάλη προσέγγιση, ε, όπως ε, είπα ε, και στη συνάδελφο και φίλη Βίκστρομ. Υπάρχουν έννοιες οι οποίες δημιουργούν ακόμη πρόβλημα Υπάρχουν διαφορετικέ θέσει ε, στο Συμβούλιο από αυτή που έχουμε θέτησει εμεί στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει όμω πολύ καλή θέληση, ε, τουλάχιστον από πλευρά τη Δανέζική Προεδρίας. Κάποια στιγμή υπήρξε κάποια μεγαλύτερη προσέγγιση. Αναγνωρίζουν όμω και οι ίδιοι οι Δανείοι ότι δεν έχουν επαρκή εντολή. Από τη στιγμή που δεν έχουν λοιπόν επαρκή εντολή και αφού στην προσεχή συνεδρίαση δεν θα την έχουν την εντολή αυτό, αυτή, γιατί δεν θα υπάρξει συνεδρίαση του Κορεπέρι ή του ε, Συμβουλίου. Είναι κάπως ασταθής ε, ακόμη η κατάσταση. Ναι, μεν υπάρχει καλή βούληση, υπάρχει έτσι μια αίσθηση ότι υπάρχει διάθεση για προσέγγιση, αλλά υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες που σας προανέφερα. Υπάρχουν τώρα κάποια προβλήματα. Εμείς ε, βασιζόμαστε σε αυτά που περιλαμβάνονται στους ορισμούς, που είναι και θέματα της δικής μας αρμοδιότητας. Έχουμε σημειώσει πρόοδο και σε κάποιους ορισμούς του πακέτου αυτού για το άσυλο. Γιατί επαναλαμβάνω ότι πήραμε τους ορισμούς, παραδείγματος χάρη για την οικογένεια και κάποιους άλλους ορισμούς. Ωστόσο, θέλουμε να είμαστε συνεπείς και με αυτά που συμφώνησαν οι συνάδελφοί μας σε άλλα θέματα. Ποιο είναι τώρα το πρόβλημα, ότι οι ίδιοι δεν συμφωνούν, παρότι εμείς συμφωνήσαμε τους Δάνους σε αυτά τα σημεία, δεν συμφωνούν με πράγματα που έχουν κλείσει ε, σε άλλους τομείς, σε άλλους φακέλους. Θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσετε κι εσείς, ε, κύριε Πρόεδρε, να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέπεια και συνεκτικότητα στο πακέτο αυτό. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει και εμένα στην Επιτροπή Γιούρι, λεγόμενος Better Regulation. Better Regulation, συγγνώμη, καλύτερη, το, το εφνομοθετήν. Και με τη Δανέζικη Προεδρία υπάρχουν πράγματα με τα οποία έχουμε συμφωνήσει, είναι ήδη κλεισμένα, έχουν κλειδώσει όπως λέμε Το θέμα είναι να ολοκληρώσουμε και τους ορισμούς ε, και κάποιες ε, νομικές έννοιες για το legal custody, παραδείγματο χάρη, και άλλους ε, ορισμούς και έννοιες. Πρέπει να γίνουν αποδεχτές. Ελπίζουμε να υπάρξει πράγματι προσέγγιση στα σημασιολογικά και νομικά ζητήματα, αλλά υπάρχουν και άλλες ε, διαφορές για την ε, δωρεάν νομική συνδρομή, παραδείγματο χάρη, κάποια θέματα σχετικά με την κράτηση. Πρόσβαση στην αγορά εργασία. Εγώ συμφωνώ με τον Επίτροπο Μάλμστρομ. Αν εδώ δεν επιτευχθεί πρόοδος και αν δεν έχουμε κάτι καλύτερο σε σχέση με αυτό που έχουμε σήμερα δεν μπορούμε να κλείσουμε με αυτήν την ε, οδηγία. Αναγνωρίζω βέβαια ότι είναι δύσκολη θέση της Προεδρίας. Γιατί πολλές χώρες βρίσκονται μέσω προεκλογικής εκστρατείας και τους ενδιαφέρει πώς θα μπορούσαν να ερμηνευθούν από τρίτους κάποια πράγματα. Η επίτροπο Μάλμστρομ τα έχει πει πάρα πολύ καλά και εμείς τα έχουμε αναλύσει και στην Επιτροπή Λίμπε. Δεν θέλουμε όμως ε, να κάνουμε πράγματα για το Θεαθήνε ουσιαστικά. Θέλουμε να μειώσουμε το κόστος για όλες τις χώρες. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο για τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν αυτά τα θέματα λοιπόν και κάποια άλλα που δεν έχουν ακόμη κλειδώσει, αλλά όπου να είναι θα ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση. Επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε και τη δική σας βοήθεια και διαμεσολάβηση, ώστε τουλάχιστον στην προσεχή συνεδρίαση να μπορέσει να δεχθεί και η Δανέζικη Προεδρία. Τις έννοιες που έχουν ήδη γίνει δεκτές. Ορισμοί που έχουν ήδη γίνει δεκτοί, γιατί επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν άλλες οδηγίες στο ίδιο όμως το πακέτο και εκεί έχουν γίνει δεκτοί κάποιοι ορισμοί, κάποια θέματα έχουν κλείσει. Πρώτα, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, ενημέρωσή σας κύριε Μασίπης ότι αφορά ε, τη, τον τριμερή διάλογο και το πώς εξελίσσεται. Θα ζητήσουμε πράγματι για μια ακόμη φορά και εμείς από το Συμβούλιο ότι η Δανική Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο ε, ουσίας της διάταξης. Προτού όμως περάσουμε σε αυτό θα ήθελα να σας πω ότι υπάρχει ένα τηλεοπτικό συνεργείο το οποίο ζήτησε να το επιτραπεί να πάρει κάποιες εικόνες των συζητήσεών μας για, για το πακέτο της ε, προστασίας δεδομένων. Πρόκειται για το τηλεοπτικό συνεδρίο Atomos Film West. Και θα περιληφθούν αυτές οι εικόνες σε ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θα γυρίσουν. Λοιπόν, περνάμε τώρα στην ε, Έκθεση «Χάνονται ζωέ στη Μεσόγειο θάλασσα. ποιο είναι υπεύθυνο της επιτροπή μετανάστευση Προσφύγων και Εκτοπιστέντων από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχουμε εδώ την εισηγήτρια τη κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, την κυρία Τίνε Κεστρίκ, ενώ είναι παρόν και ο πρόεδρος της Επιτροπής Μετανάστευσης, ο κύριο Τζάκομο Σαντίν. Σα καλωσορίζουμε θερμότατα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και με πολύ μεγάλη χαρά συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο τη Ευρώπη και την Κοινοβουλευτική του Συνέλευση, ιδίω δε σε αυτό το τόσο λεπτό θέμα ε, πολιτικών που έχουν να κάνουν με ολόκληρη την Ευρώπη. Α ακούσουμε πρώτα την κυρία Στρίκ θα έλεγα να μην περιβείτε, κυρία Στρίκ τα 10 λεπτά. Και μετά θα δώσω το λόγο στον κύριο Σαντίνη, εφόσον επιθυμεί να κάνει κάποιες παρατηρήσεις πριν από την άρξη της συζήτησης. Κυρία Στρίκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και από την πλευρά μου εσάς που μας καλέσατε εδώ να παρουσιάσουμε την εκθεσία αυτή. Είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό το να υπάρχει συνεργασία των επιτροπών μας και θα μπορούσαμε έτσι να είμαστε και συμπληρωματικοί και πιο αποτελεσματικοί. Η έκθεσή μου έχει να κάνει με τα τραγικά συμβάντα που συνέβησαν πριν από 14 μήνες όταν 63 ε, άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Μεσόγειο. Πολλές ε, αρχές βέβαια γνώριζαν πού βρίσκονταν αυτά τα άτομα και ήξεραν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ε, βρίσκονται σε δύσκολη κατάσταση και χρειάζονται βοήθεια. Θα ήθελα, επειδή δεν είναι πολύ ο χρόνο που έχουμε στη θέση μα να σα παρουσιάσω συνοπτικά τα συμβάντα. Μετά θα σα εκθέσω τα πορίσματα τη έκθεσής μου, ποιε είναι οι συστάσει στι οποίε διατυπώνω και βέβαια θα ήθελα να επιστήσω και την προσοχή σας ε, στις ε, υποδείξεις που ε, θέλω να απευθύνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε προ αυτήν την κατεύθυνση, Πώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να δώσει μια συνέχεια σε αυτή την έκθεση. Εν συντομία λοιπόν, τι έγινε με το συγκεκριμένο συμβάν το οποίο εγώ αξιολόγησα. Έχει να κάνει συγκεκριμένα με 72 άτομα από την Ποσαχάριο Αφρική που έφυγαν από τη Λιβύη λόγω της ένοπλης ε, ε, σύρεξε ένα σκάφος 7 μέτρων. Ήταν υπερφορτωμένο το σκάφος αυτό. Ουσιαστικά ο ένας καθόταν, ήταν στιβαγμένος πάνω στον άλλον, άνθρωποι αυτοί, ε, γιατί το παραφόρτωσαν οι ε, σωματέμποροι ε, και πολύ μετά από την, τον απόπλου τους από την Λιβύη αντιμετώπισαν προβλήματα, υπήρχαν και πολλά παιδιά. Μετά από 18 ώρες ε, ε, ζήτησαν βοήθεια. Υπήρξε αντίδραση και από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στην Νάπολη. Ε, εντοπίστηκε η θέση τους, το στίγμα τους και παρόλα αυτά 63 άτομα από την πείνα, την δίψα πέθαναν ενώ 11 ε, κατάφεραν μετά από 15 ε, ημέρες ε, που ήταν στη Μεσόγειο, στα νερά στη Μεσόγειο, να φτάσουν πάλι πίσω στις ακτές της Λιβύης. Δεν είναι η μόνη ιστορία αυτή, το μοναδικό τέτοιο περιστατικό. Ξέρουμε ότι τουλάχιστον 1.500 άτομα έχασαν τη ζωή τους το 2011 στην Μεσόγειο. Και είναι μοναδική περίπτωση αυτή γιατί εδώ έχουμε επιζώντες και μπορούμε να τους ζητήσουμε να μας πούν τι έγινε. Είχαμε δηλαδή καταθέσεις, ακούσαμε επίσης καταθέσεις ε, ατόμων που επέβαιναν σε σκάφη τα οποία ε, έσπευσαν στην περιοχή. Είναι νομίζω πολύ χρήσιμο αυτό γιατί έτσι μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συνέβη αυτές τις 15 μέρες και να δούμε τι διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε για να αποτρέψουμε ε, την επανάληψη τέτοιου, τέτοιων τραγικών φαινομένων το ναυτικό κέντρο της Ρώμης ε, έκανε μία κλίση έκτακτης ανάγκης για βοήθεια και στο κέντρο της Νάπολης ε, αλλά και στα σκάφη. Αλλά η Νάπολη δεν μπορούσε, ε, τα στρατιωτικά σκάφη που ήταν εκεί δεν μπορούσαν να... γιατί ήταν εμπιστευτικές οι πληροφορίες δεν μπορούσε να εντοπίσει το στίγμα. Πάντω υπήρχε επικοινωνία με τις ταλικές ναυτικές αρχές που μπόρεσαν και τους έδωσαν το στίγμα και το ακριβές αυτών των στρατικών πλοίων και από αυτή την επικοινωνία έμαθαν ότι υπήρχε μια ισπανική φρεγάτα 11 μίλια από το, σε απόσταση από αυτό το το σκάφος με το πρόβλημα και 37 ε, μίλια από το ίδιο σκάφος υπήρχε και ένα Ιταλικό ε, σκάφος. Ήταν ε, πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς τι πλοία είναι κοντά στην περιοχή, ποια είχαν τη δυνατότητα, είχαν πάνω τους ελικόπτερα. Γιατί αφού δόθηκε ο συναγερμός μπορούσαν τα ελικόπτερα αυτά να υπερίπτανται πάνω από το σκάφος δίνοντας κάποια εμφάρυνση λέγοντας στους ανθρώπους αυτούς μείνετε εκεί που είστε, τους ε, πέταξαν και κάποια τρόφιμα, νερό και τους είπαν ότι θα έρθουν να τους ε, ε, σώσουν. Και πραγματικά αυτό μας είπαν και οι διασώστες και τα άτομα είχαν εμπιστοσύνη, ήξεραν ότι θα σώθουν. Τελικά όμως όχι, δεν γύρισε κανένας. Και μετά ήρθαν άλλα δύο ψαράδικα πολύ κοντά στο σκάφος αυτό είχαν επαφή με τα άτομα, με χειρονομίες, με κινήσεις, ε, αλλά και προφορικά μπόρεσαν να έχουν κάποια επικοινωνία, αλλά και αυτά τα ψαράδικα εγκατέλειψαν το σημείο και δεν ξανάρθαν. Δέκα μέρες μετά, αφού πια είχαν πεθάνει ήδη πάνω στο σκάφος, ήρθε ε, ένα μεγάλο σκάφος που είχε και ελικόπτερο πάνω ε, και πάνω στο κατάστρωμα υπήρχαν άνθρωποι με στρατιωτικέ στολέ, κοιτούσαν με τα γυάλια, φωτογράφησαν τους ανθρώπους αυτούς. Και αυτοί όμως αποφάσισαν να, να φύγουν, να αποπλέψουν μακριά, αφήνοντας αυτούς τους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν αυτά τα προβλήματα. Θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε τελικά πού ήταν αυτά τα στρατιωτικά πλοία, να ξέρουμε τη θέση του στην ακριβή. Και θέλουμε να ξέρουμε και ουσιαστικά να έχουμε πρόσβαση και στο ημερολόγιο ε, του, του πλοίου. Τι έκαναν ε, τα ελικόπτερα. Είχαν κάποια συμμετοχή. Τι πώς κινούνταν, τι έκαναν τα ελικόπτερα και τα σκάφη. Έγιναν, ε, έλαβαν μηνύματα, τα μηνύματα αυτά από την Άπολη, ε, από τον ΝΑΤΟ δηλαδή και από τη Ρώμη ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονταν βοήθεια. Εμείς ζητήσαμε από όλους ε, όσους βρίσκονταν εκεί στην περιοχή να δώσουν πληροφορίες ή να βρουν πληροφορίες. σε σχέση με αυτό το συμβάν και περιμένουμε ακόμη συγκεκριμένες απαντήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Γαλλία, γιατί υπήρχε ένα τηλεκατευθυνόμενο ε, σκάφος από τη Γαλλία, το οποίο έλαβε μια φωτογραφία, πήρε μια φωτογραφία του σκάφους πριν όμως ε, ε, προκύψουν τα προβλήματα και το έστειλε στο κέντρο συντονισμού. Αλλά η Γαλλία ακόμη δεν μας έχει δώσει απάντηση για το προκείμενο συμβάν. Θέλουμε επίση να έχουμε και από την Ισπανία περισσότερα στοιχεία, γιατί υπήρχε πολύ κοντά το, σπίτι, το σκάφο Μέντεθ Νούνιεθ, αυτή η φρεγάτα. Αυτοί λένε όχι, ε, δεν μας ενημέρωσαν, ούτε ήμασταν 11 μίλια μακριά. Δεν μας είπαν όμως πού ακριβώς ήταν, ποια ήταν η θέση του σκάφους αυτού. Δεν ήταν 11 μίλια, πόσο ήταν. Το ΝΑΤΟ ταυτόχρονα μας λέει ότι ήταν ενημερωμένα όλα τα πολεμικά σκάφη και η Ισπανική φρεγάτα επομένω ήταν ενημερωμένη. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις σε πληροφορίες που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη και από τις πληροφορίες που έχουμε πάρει από τον ΝΑΤΟ δεν έχουμε βγάλει σαφή εικόνα. Θέλουμε λοιπόν να ξεκαθαρίσει κατάσταση, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, πού βρίσκονταν τα σκάφη. Αυτό το ελικόπτερο ε, που, ήταν πάνω από που πέταξε πάνω από το σκάφος και αυτό μεγάλο πολεμικό που προσέγγισε ποιες, από ποιες χώρες ήταν. Και θέλουμε και από τα Υπουργεία Άμυνας των χωρών να έχουμε πληροφορίες. Τελικά με όλα αυτά που κάναμε καταλήξαμε ε, στο ότι δεν υπάρχει μία και μόνη ε, αρχή που να είναι ε, υπεύθυνη. Ουσιαστικά πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν ό,τι έπρεπε Υπήρχαν πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαν σε πολλές περιπτώσεις να είχαν βοηθήσει ε, αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα οι σωματέμποροι αυτοί που πραγματικά δίστακτα ε, φόρτωσαν όλους αυτούς τους, στίβαξαν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτοί έχουν μέρη δύο ε, πολύ σημαντικό. Ούτε και οι αρχές όμως ε, έκαναν ε, ε, αυτό που έπρεπε όταν πλέον αντιμετώπισε δυσκολίες αυτό το, το μικρό πλεούμενο στο οποίο ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Ούτε τη συντονισμένη ευθύνη ανέλαβαν από το κέντρο ώστε να υπάρξει μια συγκεκριμένη δράση διάσωσης. Υπάρχει μια κατευθυντήρια γραμμή από τον Διεθνή Οργανισμό, τον IMO, που λέει ότι το κράτος που θα πάρει το πρώτη, την πρώτη κλίση πρέπει να λάβει την ευθύνη μέχρι σότου αναλάβει την ευθύνη το κράτος το οποίο ε, βρίσκεται η σωστική ζώνη κατά κάποιο τρόπο. Εμείς δεν μπορούσαμε να συντονίσουμε ε, έτσι θεωρεί και το ΝΑΤΟ. Πρέπει να, να γίνει μια περαιτέρω διερεύνηση, αλλά και το ΝΑΤΟ ε, από ό,τι φαίνεται υπήρχαν πολλά σκάφη υπό τη δίκηση του ΝΑΤΟ εκεί στην περιοχή. Σίγουρα ε, θα πρέπει να τηρούν τις διεθνείς δεσμεύσεις τα κράτη, αλλά και το ΝΑΤΟ έχει έναν ρόλο συντονισμού. ώστε να εξασφαλίσει τη τήρηση των εθνών υποχρεώσεων των κρατών. Ιδίω ε, τώρα, λοιπόν, με αυτή την έρευνα ε, και εμεί έχουμε καταλήξει ω μπέρασμα ότι θα πρέπει να συνεργαστεί πλήρω μαζί μα το ΝΑΤΟ και να μα δώσει πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία που χρειαζόμαστε για να βρούμε του υπεύθυνου. Υπήρχαν και κάποιες άλλες διαφωνίες σε σχέση και με το ναυτιλιακό δίκαιο. Μας λέει το ΝΑΤΟ ότι τα μηνύματα δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα Δηλαδή ήταν ε, μια κλίση εκτακτής ανάγκης, ε, ήταν ένα distress call. Ε, στην Ιταλία έχουν ξεκάθαρους ορισμούς. για το αν πρόκειται για σήμα κινδύνου, για κατάσταση εκτακτής ανάγκης. το distress, το σήμα κινδύνου είναι ξεκάθαρο ουσιαστικά. ενώ είναι ξεκάθαρο πώς δεν αντιδρά κανείς. Δεν θα πρέπει αυτές οι έννοιες ε, να έχουν μια συνεκτική αντιμετώπιση κοινή από όλους. Επίσης το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι δεν συνεργάστηκε πλήρως ε, και με τις ε, Ιταλούς συνοριοφύλακες, border guards. Φυσικά και ξέρουμε, ξέραμε για την περίπτωση εκείνη της Λιβύης ότι πάρα πολλοί θα μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα. Έπρεπε να υπάρξει μια συνεργασία με τους αεροφύλακες για να είναι ξεκάθαρο ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για ποια δράση. Για να μην δημιουργηθεί περισσότερο χάος τελικά, ούτε να προκύψουν διαφωνίες. Πρέπει να υπάρχει συντονισμένη δράση σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν πρέπει να χαθεί καμία ζωή ανθρώπινη. Τώρα, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανέφερα δύο συγκεκριμένες συστάσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλω να μπω σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες θεμάτων που θα πρέπει να παρακολουθήσετε. Καταρχάς, να βρεθεί να καταλάβετε τι ακριβώς συνέβη. Χρειαζόμαστε δορυφορικές πληροφορίες, ούτως ώστε να καταλάβουμε και εμείς οι ίδιοι εάν η θέση όλων αυτών των στρατιωτικών σκαφών ήταν γνωστή. Ποια ήταν αυτή η θέση. Ούτε τα κράτη-μέλη, ούτε η Βαρόνια Άστον μας έδωσε πρόσβαση σε δορυφορικές πληροφορίες. Τότε μας είπε ότι δεν υπήρχαν καθόλου ε, δορυφορικές πληροφορίες για τη Μεσόγειο, γιατί υποτίθεται ότι εστιαζόταν στα σύνορα με την Τινησία για να αντιμετωπίσουν το ανθρωπιστικό πρόβλημα. Επομένως δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά δορυφορικά στοιχεία. Μας παρέπεμψε στο ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ φυσικά είπε ότι δεν έχει καθόλου πληροφορίες δορυφορικές για την περιοχή. Πολύ περίεργο μου φαίνεται, γιατί αν υπάρχει μια στρατιωτική επιχείρηση εν εξελίξη, κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν δορυφορικές πληροφορίες για την περιοχή. Βρήκαμε όμως ότι Υπάρχουν υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δορυφορικέ πληροφορίες για την περιοχή και μάθαμε ότι η Φερρυπίν, το κοινό ερευνητικό κέντρο, ασχολείται με την ανείχνευση των σκαφών, με τον εντοπισμό των σκαφών. Μπορείτε να ζητήσετε λοιπόν από αυτούς να σας δώσει πρόσβαση σε αυτές τις δορυφορικές πληροφορίε. Το ίδιο ισχύει και για δύο οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα λίας, την ΕΦΚΑ και την ΕΚΑ, που είναι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν τέτοιες πληροφορίες δορυφορικές. Κάτι άλλο που έχω ήδη πει. Μπορείτε να πάτε στα Υπουργεία σας, τα εθνικά, ούτω ώστε να μας δώσουν αυτά τα Υπουργεία τις πληροφορίες για τη θέση των σκαφών και κάτι ακόμα. Υπάρχουν κάποια νομικά κενά. Βρήκαμε τρία βασικά νομικά κενά. Καταρχάς, οι ευθύνε. Υπάρχει μια φαιά ζώνη που δεν καλύπτεται αυτή τη στιγμή ο IMO και η Ιταλία διαφωνούν. Αυτές οι διαφωνίες θα πρέπει να επιληθούν. Επίσης, η διαφωνία για την κάθοδο από το σκάφος. Αλλιώς ερμηνεύει, ερμηνεύει η Μάλτα για το ποιος είναι υπεύθυνο για την αποβίβαση και αλλιώς άλλα κράτη-μέλη. Ποιος είναι υπεύθυνο για την αποβίβαση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί δεν ασχολούμαστε μόνο με έρευνα και διάσωση, αλλά υπάρχει μια ολόκληρη αλυσίδα εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές μετά τη διάσωση ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη. Ποιος παίρνει αυτούς τους ανθρώπους, ε, τους αποβιβάζει, ποιος τους δίνει πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, ποιος τους δίνει, τους εξασφαλίζει εγκαταστάσεις. Ε, μπορεί να υπάρχουν απροθυμίες για τη διάσωση. Ας πούμε αυτά τα εμπορικά σκάφη, ας πούμε, ε, μπορεί να, είναι, να διστάζουν ε, να αποβιβάσουν αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά και τα κράτη που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του μετόπου και που φέρουν το μεγαλύτερο βάρος. Θα πρέπει να ασχοληθούν αυτά κυρίως με όλους τους μετανάστες ε, μετά τη διάσωση. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι και άλλα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να δείχνουν αλληλεγγύη και πρέπει να μοιραστούν αυτή την ε, ευθύνη. Ε, υπάρχει θέμα με την κατάσταση των μεταναστών. Ε, Ποιο θα δώσει τους πόρους. Όλα αυτά τα θέματα είναι προς συζήτηση. Και αν επιληθούν θα βοηθήσουμε τη διαδικασία διάσωσης αυτή αυτή. Επίσης το δίκαιο της θάλασσας δεν είναι ευρωπαϊκό δίκαιο, είναι μία ε, ένα διεθνές δίκαιο, τμήμα του διεθνούς δικαίου. Αλλά μπορεί να συνεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και να βρεθεί μια κοινή θέση για την τροποποίηση αυτών των συμβάσεων, ούτω ώστε ε, να είναι δεσμευτικέ. Και το τελευταίο σημείο που θέλω να θέσω εδώ, κάνουμε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα δεσμευτικό πρωτόκολλο για τη Μεσόγειο και να ασχολείται αυτό το πρωτόκολλο με όλα τα θέματα που αφορούν την Μεσόγειο και αντιμετωπίζει το πρόβλημα των ανθρώπων που δεν διασώζονται. Ε, αποβίβαση, μετεγκατάσταση. Όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να επιληθούν στα πλαίσια μίας και μόνης επιχείρησης. Υπάρχει επιμερισμό τη ευθύνη. Αυτό είναι δεδομένο. Και δεν θα πρέπει να αφήσουμε μόνοι του κάποια κράτη-μέλη που τυχαίνει, εν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρό και να αντιμετωπίζουν πρώτα αυτά τα προβλήματα. Πολύ λεπτομερή η έκθεση. Να ανοίξουμε λοιπόν ε, τη συζήτηση. Ο κύριος Αντένη ίσως θα ήθελε να προσθέσει κάποια σχόλια, αν το επιθυμείτε. Σας παρακαλώ εν συντομία για να διατηρήσουμε και τον ε, χρόνο ομιλίας. Στο γνωρίζω τους κανόνες του Κοινοβουλίου, γιατί πριν γίνω ε, γερουσιαστής στην Ιταλία ήμουνα 10 χρόνια ευρωβουλευτής. Ε, ευχαριστώ λοιπόν και χαιρετίζω όλους εδώ τους συναδέλφους. Είμαι πολύ ικανοποιημένος που έρχομαι εδώ και μπορώ να σας μιλήσω για τις δικές μας εμπειρίες για να σας πω ε, τι κοινέ εμπειρίες έχουμε εμεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρώπης, που δεν είναι ε, αντιφατικές αλλά συμπληρωματικέ. Επειδή υπήρξα και τα δύο, σας λέω ότι στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχει η δυνατότητα να ψάξουμε αυτά τα θέματα. Υπάρχουμε, έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να παρέμβουμε, για να ολοκληρώσουμε δηλαδή τις δράσεις μας. Ε, και ακριβώ αυτό ζητάει η συνάδελφο που μίλησε πριν, με αυτή τη φανταστική παρουσίαση που έκανε. Ε, βοηθήστε μα. Βοηθήστε μα να υπάρξει μια συνέχεια σε αυτό το πρόβλημα. Βοηθήστε μα ούτως ώστε να ξεκαθαρίσουμε τι ακριβώ έγινε. Υπάρχουν πολλέ φαίε περιοχε ε, Σα Σας ε, υπενθύμησε τα γεγονότα η συνάδελφο και εντοπίστηκαν τρία επίπεδα ευθύνη. Γιατί ο τίτλο είναι Ποιο είναι ένοχο, Ποιο είναι υπεύθυνο. Ιταλία, Ισπανία και ΝΑΤΟ. Έτσι, Ιταλία. Γιατί από εκεί ξεκίνησε ε, το σήμα κινδύνου. Ο ένας από τους πρόσφυγες είχε τον αριθμό του κινητού ενός ε, ε, παπά Ερυθρέου που ήταν στη Ρώμη. Από εκεί έφυγε το σήμα κινδύνου. Ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία στη θάλασσα, όλα αυτά σωστά, αλλά υπήρξε κάποιο πρόβλημα επικοινωνία, πιστεύουμε. Ίσως κάποιος δεν πήρε σοβαρά την ιστορία αυτή. Αυτό το σήμα κινδύνου δεν έφτασε στο σωστό παραλήπτη. Δεν έφτασε εκεί που έπρεπε να φτάσει. Όταν συζητήσαμε το θέμα αυτό τον Απρίλιο ε, στο Στρασβούργο, έχουμε ένα πρόεδρο τη Επιτροπή και σα μεταφέρω το κλίμα τη ε, Συνόδου. Ε, οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Μαλτέζοι μίλησαν, πήραν το λόγο σε αυτή τη συζήτηση για να ξεκαθαρίσουν ποιο είχε την ευθύνη. υπήρχε η εθνική ευθύνη και πάνω από αυτούς υπήρχε και η ευθύνη του ΝΑΤΟ. Να σας υπενθυμίσω ότι είμαστε στο, το Μάρτιο, 26 Μαρτίου του 2011. Τότε έφυγε το ντίνγκι αυτό, το βαρκάκι. Είχαμε πόλεμο στη Λιβύη και όλη η ζώνη γύρω από τη Λιβύη ήταν πολεμική περιοχή που τη διαχειριζόταν το ΝΑΤΟ. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να μετακινηθεί κανείς με τα κλασικά σκάφη ας πούμε. Ε, όπως είπε και η συνάδελφος, το ΝΑΤΟ έχει τα δικά του σκάφη και σε κέρυε θέσει ούτως ώστε να καταλάβει ε, τι γινόταν στην περιοχή. Ήξερε πολύ καλά για αυτό τον Τίνκι. Ε, το ΝΑΤΟ, ε, σε μια συζήτηση που είχαμε στο Βουλίο τη Ευρώπης, ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Εγώ ως πρόεδρος της Καθήλυνα Αρμόδιας Επιτροπής αρνήθηκε πάρα πολλά πράγματα. Προφανώς, οι μαρτυρίες των επιζώντων μας λένε πολλά, μας ξεκαθαρίζουν πολλά, αλλά το ΝΑΤΟ αρνείται το σύνολο της μαρτυρίας, δεν τα δέχεται όλα αυτά τα στοιχεία. Εμείς θέλουμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα να διευκρινιστούν για να βγει και να λάμψει η αλήθεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ψαράδικα αυτά, που πλησίασε αυτούς απελπισμένους ας πούμε και δεν τους βοήθησε, τώρα εδώ υπάρχει μια εκδοχή. Μπορεί, α πούμε, οι ψαράδες αυτοί να φοβούνταν να έρθουν σε επαφή με αυτά τα σκαφίδια. Το έχουμε συζητήσει και στην Λαμπεντούζα σε μια επίσκεψη που κάναμε. Γιατί μπορεί λένε, μας λένε τώρα αυτοί, να μπουν σε μια δικαστική περιπέτεια, ας πούμε. Μπορεί να θεωρηθεί ότι διευκολύνουν, ας πούμε, τη αυτομετανάστευση. Και όχι μόνο αυτό. Συχνά από αυτές ε, τις βάρκες των ε, απελπισμένων ε, προκύπτουν άνθρωποι με κακές ε, προθέσεις και καμιά φορά, ας πούμε, μπορεί να πάγουν και τους ψαράδες. Είναι απίστευτο το ότι δεν πλησίασε κανένα ψαράδικο. Επίσης έχουμε την ακτοφυλακή, έχουμε τους καραμπινιέρους, ε, τους επαγγελματίες εν πάση της διάσωσης. Κανονικά ε, πρέπει να πλησιάζουν ε, από πολλά σημεία ένα τέτοιο σκαφίδιο ας πούμε, για να το σώσουν. Πάντως εμείς εγκρίναμε την έκθεσή μας με μεγάλη πλειοψηφία στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχουν κάποια σκοτεινά σημεία που πρέπει να ξεκαθαριστούν, αλλά σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε το θέμα. Επίσης, ξέρουμε ότι αν υπάρχει ένας ευθύνης, ε, υπεύθυνος, συγγνώμη, είναι η Λιβύη. Αλλά εκείνη τη στιγμή η Λιβύη δεν υπήρχε, γιατί ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Και ακόμα και δύσκολο, ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να πάμε στους Λίβιους, τους που είναι υπεύθυνοι, ας πούμε, και να ζητήσουμε ευθύνες. Αυτοί οι άνθρωποι 18 μέρες έπλεαν απελπισμένοι στη θάλασσα. Το σκάφο τελικά επέστρεψε στη Λιβύη, στις ακτές της Λιβύης. Αλλά ε, δεν είχε όλα τα άτομα, δεν είχε δηλαδή και τα 72 άτομα. 62 ε, ήταν οι νεκροί, 10 οι επιζώντες, ο ένας από αυτούς πέθανε α, γιατί ήταν σε κακή κατάσταση, 9 τελικά σώθηκαν. Εμείς συζητάμε αυτά τα, τα πράγματα. Ε, στη Λαμπεντούζα εντωμεταξύ αντιμετωπίζουμε συνέχεια τέτοια προβλήματα. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται. Μέσα σε 20 χρόνια χιλιάδες άτομα πέθαναν στη θάλασσα. Πάνω από 100.000 έχουν αποβιβαστεί. Αυτό το θέμα πρέπει να το ψάξουμε στο μέλλον. Δεν πρέπει να κάνουμε κι άλλα τέτοια λάθη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαντίνη δεν παίρνει το λόγο για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο. Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε που ήρθε και να του ευχηθούμε καλή επιστροφή στη Συμβούλιο της Ευρώπης. Μάλιστα, να έχετε υπόψη σας πριν ξεκινήσετε, γιατί ο κατάλογος των ομιλητών είναι πολύ μακρύς. Δέκα μέλη τουλάχιστον ε, περιλαμβάνει και ο κύριο Μπρόντς. Δύο λεπτά σας παρακαλώ πολύ. Ιδάλλως δεν θα καταφέρουμε να τηρήσουμε το χρονικό όριο προκειμένου να ολοκληρώσουμε την συνεδρίαση μέχρι τις 6 και 4. Σας παρακαλώ λοιπόν δύο λεπτά. Ο κύριος Μπουζουτήλη έχει το λόγο καταρχάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους δύο εκπροσώπους του ΠΙΕΣΗ για την παρουσίασή τους και για τα συμπεράσματα που εξαγάγαν. Και οι δύο αυτό που επισημαίνουν είναι ότι ουσιαστικά το μοναδικό συμπέρασμα είναι ότι θα πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη. Τρία συμπεράσματα. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα πριν από 14 μήνες. Τους τελευταίους 14 μήνες έχουν εμφανιστεί παρόμοια περιστατικά. Εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη θάλασσα και αυτό εξακολουθεί να συμβαίνει εδώ, την ώρα που μιλάμε. 500 άτομα διάσωσε η χώρα μου στη θάλασσα τον τελευταίο μήνα και μιλάμε για μια μικρή χώρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός των ατόμων που διασώστηκαν. Και σε κάθε περίπτωση σχεδόν αυτοί που διασώθησαν δηλώνουν ότι κάποιοι άλλοι χάθηκαν στη θάλασσα. Καλό λοιπόν είναι να ερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά ποτέ να μην ξεχνάμε ότι το θέμα είναι πώς θα πρέπει να γίνει η πρόληψη για να μην ξανασυμβούν τέτοια πράγματα, γιατί συμβαίνουν κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά τους, ε, τα άτομα που κάνουν αυτή την λαθρέα ε, μεταφορά των ατόμων αυτών. Αυτοί είναι οι πραγματικοί εγκληματίες, γιατί οργανώνονται μέσω εγκληματικών ε, κυκλωμάτων και γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά για κανέναν άλλο λόγο. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να εκδοθούν αυτοί οι λαθρέμποροι ανθρώπων, όπως ζητούμε να εκδίδονται και οι πειρατές ε, της Σομαλίας. Αυτό κάνουμε με τους πειρατές της Σομαλίας, γιατί να μην το κάνουμε αυτό και με τους ε, λαθρεμπόρους ε, που μετακινούν λαθρέα άτομα στην Μεσόγειο. Και τέλος, κάποιος ε, θα πρέπει να λάβει την ευθύνη. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ποιος τους σώζει αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι ποιος θα τους αναλάβει μετά την αποβίβασή τους. Και αυτό δεν το θίγουμε γιατί κανείς δεν θέλει να μοιραστεί την ευθύνη. Άρα, μέχρι ότου όλοι αποτεχτούμε ότι θα πρέπει να μοιραστούμε την ευθύνη αυτή, δυστυχώς θα πρέπει να υπάρχει υπεραιτέρω ε, διάλογος. Ευχαριστώ, κυρία ε, Ρομέρο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το Συμβούλιο της Ευρώπης που ερευνά τα ζητήματα αυτά. Είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Αλλά, όπως είπατε, δεν είναι μονομένο περιστατικό αυτό που εμφανίστηκε να σας πω ότι και στο Ισπανικό Κοινοβούλιο στη δεκαετία του 80 είδα ναυάγια σε διάφορες περιοχές και σε όλα αυτά τα χρόνια καλούσα την Ισπανική κυβέρνηση να επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Μία από τις λύσεις που πρότεινε η Ισπανική κυβέρνηση είναι κοινέ περιπολίες. Με συμμετοχή δηλαδή Ισπανίας και Μαρόκου που στην προκειμένη περίπτωση ήταν η χώρα από την οποία έφευγαν μετανάστες. Αυτές οι κοινέ περιπολίες ήταν μια πραγματική καινοτομία και πολύ επιτυχημένη λύση που επέτρεψε να υπάρξει έλεγχος στα ναυάγια αυτά. Και υπάρχει ένα πρωτόκολλο πλέον για τα ναυάγια αυτά. Αλλά ε, γι' αυτό θεωρώ πόσο, ότι είναι σημαντικά σημαντικές εντιμερείς συμφωνίες αυτές. Μιλάμε για την ε, ναυτική προστασία και ασφάλεια. Για την ασφάλεια στη θάλασσα. Πρέπει να υπάρξει κοινή δράση. Η Αταλάντη είναι μια επιχείρηση που αποτελεί ένα παράδειγμα τέτοιας κοινή δράση και νομίζω ότι και το Γραφείο Ασύλου της Μάλτας ε, κάπου ε, πρέπει να εξυπηρετήσει και εξυπηρετεί προς αυτή την κατεύθυνση μεταξύ άλλων. Είναι τόσες πολλές αυτές οι περιπτώσεις ε, σχεδιών και άλλων ε, μικρών πληγούμενων που ναυαγούν Πρέπει να βρούμε βέβαια ευθύνε. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν από πολέμους κτλ. Αλλά σίγουρα πρέπει να δοθούν εξηγήσει. Αν δεν έχει δώσει η Ισπανική κυβέρνηση επαρκή εξή, πρέπει να δώσει επαρκή εξηγήσει. Και αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει με τα κέντρα αυτά ε, και με αυτού του οργανισμού Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει πάνω το δυνατό. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτή η τραγωδία όμω δεν θα πάψει. Ε, γιατί ε, υπάρχουν πόλεμοι και θα πρέπει και οι ευρωπαϊκές υποδομές να είναι στο ύψος ε, των περιστάσεων. Και αυτό πρέπει να ισχύει και από τις δύο όχθες της Μεσογείου. Κυρία Βέμπρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους προσκεκλημένους μας για το έργο που έχουν επιτελέσει ως τώρα και για την παρουσίαση της έκθεσης αυτής. Συμφωνώ με τους συναδέλφους σε πολλά από τα ζητήματα που ανέφεραν και πρέπει να σας πω ότι ντρέπομαι βαθύτατα που μπορούν και συμβαίνουν τέτοια πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Και για διάφορους λόγους και με πολύ κινησμό αφήνουμε τον κόσμο να πεθαίνει γιατί το πρόβλημα, όπως είπατε, είναι ποιος θα τον αναλάβει μετά. Και επειδή δεν τον συμφωνούμε από αυτού, τους αφήνουμε να πεθαίνουν. Πολύ απλά. Νομίζω ότι στο ποινικό δίκαιο των κρατών μελών υπάρχουν διατάξεις που ορίζουν ότι αν ε, αφήσουμε κάποιον που υποφέρει να πεθάνει, ε, αυτό τιμωρείται με ποινική κύρωση. Εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ποιο, σε ποιο βαθμό είναι υπεύθυνο το ΝΑΤΟ. Φέρει μέρος της ευθύνης. Αλλά ως πολίτης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως μέλος της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι να κάνει. Ιδάλλως, κοιτάξτε, έχουμε δουλέψει σκληρά για όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Προσπαθούμε να παρέχουμε πιο πολύ χρηματοδότηση και τελικά τι κάνουμε, μετράμε πόσοι πέθαναν. Και για να είμαστε ειλικρινείς, κοιτάξτε, τα άτομα που έφυγαν υπό τέτοιες συνθήκες δεν ναι, έφυγαν γιατί ήθελαν να ζήσουν απλά το ευρωπαϊκό όνειρο. Όχι, έφυγαν για να σώσουν τη ζωή τους. Άρα θεωρώ ότι φέρουμε ευθύνη. Και κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Το γεγονός ότι οι λαθρέμποροι το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε, ναι, είναι οι κακοί μεν και θέλουμε να τους πιάσουμε, να τους βάλουμε στη φυλακή. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς απαλλασσόμεθα ως Ευρωπαϊκή Ένωση από την ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Αργεντίνη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ την και για την ιστορία αυτή. Όταν την διάβασα, σχεδόν σαν μυθιστόρημα ήταν το ψήφισμα αυτό και αποτελεί ένα παράδειγμα πολλών τέτοιων περιστατικών, όπως είπε ο κύριος Μπουσουτήλ, και πολλών περιστατικών τέτοιων τραγωδιών που έχουν παρουσιαστεί και στο μεταξύ. Άρα ποιος είναι υπεύθυνο και τι μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσουμε τους λαθρεμπόρους, γιατί θεωρώ ότι χρειάζεται και μία άλλη εναλλακτική μορφή πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν δεν χρειάζεται να πάρουν ε, καροδότσουφλα αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και θεωρώ ότι η πολιτική μας για το άσυλο δεν είναι σωστή και έτσι οθεί τους ανθρώπους στη λαθρέα οδό και γι' αυτό παρουσιάζονται τέτοιες τραγωδίες όπως αυτή. Κάτι διαφορετικό. Η αρνητική στάση των κρατών μελών, είτε είναι κρατημέλη μέσω του ΝΑΤΟ είτε όχι, αλλά η αρνητική του στάση για να δώσουν πληροφορίες και ανοιχτά πληροφορίες για το ποιος έκανε τι και πότε και πού. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την πολιτική για το άσυλο και πώς μπορούμε να ε, εισάγουμε τέτοιες ρητρές αλληλεγγύης όταν κοιτάμε σαν μέλη από την άλλη. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν μια τέτοια στιγμή ο κόσμος τολμάει να κοιτάει από την άλλη πλευρά, έχουμε πρόβλημα. Κύριε δύο λεπτά. Thank you, I want to thank both. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τους δύο ομιλητές, ιδιαίτερα την εισηγήτρια για την έκθεσή της, η οποία πραγματικά έκανε εξαιρετό έργο, συλλέγοντας πληροφορίες, μιλώντας με τους ε, επιβιώσαντες μιλώντας με το ΝΑΤΟ, με τις διαστοστικές δυνάμεις στη Μάλτα και το αποτέλεσμα είναι μια καλά τεκμηριωμένη έκθεση που μας ε, δείχνει με σαφή τρόπο το τι έγινε και ποιος θα πρέπει να λάβει την ευθύνη για την ε, αγνόηση του σήματος αυτό του σήματος κινδύνου. Και επίσης, να σας πω, υπάρχει και το Boats for People Project, μέσω διοργάνωσης ε, τέτοιων δραστηριοτήτων από 2 με 9 Ιουλίου θα συλλέξει ε, τέτοιες πληροφορίες για περιστατικά στη θάλασσα και αν διαπιστωθούν αποτυχίες ε, αντίδρασης σε τέτοια σωστικά μηνύματα, σήματα κινδύνου, θα υπάρξουν κυρώσεις. Θα ξεκινήσουν δικαστικές αγωγές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξουν τέτοιες να υπάρξει συνέχεια. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε την ατιμορρησία όταν ο κόσμος πνίγεται και ο κύριος Σαντίνη αναφέρθηκε στη Λαμπεντούσα αρκετές φορές και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να τονίσω πόσο σημαντικό είναι να ξανανοίξει το κέντρο υποδοχής στη Λαμπεντούσα που είχε κλείσει πριν από ένα χρόνο υπό όρους πολύ αμφισβητήσιμους. Ευχαριστώ κύριε Σαντίνη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω θερμότατα αυτή την πολύ θετική έκθεση της κυρία Στρίκ. Και θέλω να πω στον κύριο Σαντίνη ότι και εγώ διατέλεσα πρόεδρος της Επιτροπής ε, Μετανάστευσης ε, του Σύμβουλου της Ευρώπης για τρία χρόνια, άρα και εγώ ξέρω γιατί μιλάω. Η έκθεση πραγματικά αποτελεί ένα πολύ, ε, μια πολύ έντονη κλίση. Πρέπει να επιστήσουμε την προσοχή μας σε αυτά τα θέματα, αλλά θέλω να πω ότι εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη ε, στον ισπανικό στόλο και δεν πιστεύω ότι μπορεί το ναυτικό να λέει ψέματα. Η φρεγάτα Μέντεθ Νούνιεθ ή οποιαδήποτε άλλη φρεγάτα δεν υπήρχε περίπτωση να άκουγε ε, ένα σήμα κινδύνου και να μην πήγαινε να ε, επέμβει καμία επικοινωνία δεν ήρθε από το κέντρο συντονισμού διάσωσης της Ρώμης, δεν έφτασε τουλάχιστον ε, στους δέκτες ε, του, της φρεγάτας αυτής. Η φρεγάτα αυτή έδωσε επιτυχημένα βοήθεια σε δύο ε, περιπτώσεις στις 26 ε, και 27 του μήνα, σε δύο αντίστοιχες περιπτώσεις. Πώς λοιπόν παρέσχε βοήθεια σε δύο περιπτώσεις και όχι στη συγκεκριμένη δεν μπορεί ε, να υπάρχει υποψία. Πρέπει σίγουρα να διευνηθεί η υπόθεση και σε βάθος. Είναι πολύ τολμηρή αυτή η έκθεση γιατί πραγματικά ε, θέτει τον δάκτυλο από τον τύπο των ήλων. Και βάζει το δάκτυλο στην πληγή κιόλα για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομα του. Πέντε συστάσεις ε, είναι πολύ καλές οι συστάσεις και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και σίγουρα πρέπει και να ερευνήσουμε και να παληθεύσουμε όλα αυτά και πρέπει σίγουρα και να συνεργαστούμε σε αυτήν την ε, έρευνα. Τώρα, ε, η αναζήτηση των συντεταγμένων ε, των πλοίων. Καλό είναι, αλλά όταν ζητάτε για τη φρεγάτα με εντεθνή στο συγκεκριμένο χρονικό σημείο, λέτε σε ποιο χρονικό ε, σημείο ακριβώ. Είναι πολύ πλόκο. Πώ μπορεί κανεί να ε, βρει τι συντεταγμένε τόσο ξεκάθαρα. Επίση, το Μπορσίνι, ένα ιταλικό πλοίο, ήταν λέτε σε από 37 μιλίων. Αυτό πώ έχει μετρηθεί. Πρέπει να το υπολογίσουμε και αυτό ως ερώτημα. Και επίσης, πρωτόκολλο δράση στη Μεσόγειο που λέτε. Εγώ το επικροτώ και το υποστηρίζω και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Όχι όμως, κυρία μου, μόνο στην Μεσόγειο. Ρωτήστε τον πρόεδρο της Επιτροπής που ζει κοντά ε, στη, στον Ατλαντικό ε, αν εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 10.000 ε, νεκροί, εκεί στη Βόρεια Αφρική δηλαδή, στις ακτές. Το πρωτόκολλο αυτό όχι μόνο για την, μάλλον στον Ατλαντικό, που βγαίνει προς τον Ατλαντικό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να ισχύει αυτό το πρωτόκολλο μόνο για τη Μεσόλ και για τον Ατλαντικό και για παντού. Ε, ευχαριστώ. δύο λεπτά σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, θα προσπαθήσω να σεβαστώ το χρόνο. Εξάλλου, δεν θεωρώ ότι πρέπει να κάνω μεγαλόστομες δηλώσεις. Ε, θέλετε το πρωτόκολλο για το άσυλο, θέλετε να συμφωνήσουμε όλοι. Ε, όχι, εγώ θέλω να πω διαφορετικά πράγματα, δεν θέλω να συμφωνήσω με τους άλλους. Η έκθεση της κυρίας Τρίκ, τη θέλω να την ευχαριστώ. Θέλω να σε ευχαριστήσω και εσάς κύριε Σαντίνη. Αλλά είναι τόσο τρομερή τόσο παράλογη και τόσο δύσκολο να την αποδεχτούμε, που δεν μπορώ να σας πω τίποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή συζητάμε δηλαδή για εγκλήματα, για δικήματα που έχουν διαπραχθεί και για νεκρούς που πέθαναν επίτηδες. Κάποιοι φταίνε δηλαδή. Δηλαδή κάποιος δεν παρέλειψε να τους βοηθήσει. Αν εγώ ας πούμε έχω χτυπήσει κάποιον, α πούμε, με το αυτοκίνητο. Και αν δεν σταματήσω να τον βοηθήσω, πρέπει να πάω στη φυλακή, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για κανόνε. Δεν αφορούν μόνο του πολίτε, αλλά αφορούν και τι κυβερνήσει και για τα κράτη και, για... και αφορούν και τον ΝΑΤΟ. Μιλάμε για ποινικά δικήματα πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε να τα κρύψουμε πίσω από παραπετάσματα καπνού, α πούμε, ότι όλα τα κράτη είναι καλά. Καλά είναι αυτά που ακούσαμε τον Ισπανό συνάδελφο. Καλά, αλλά όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέθαναν. Ε, πρέπει λοιπόν να επιληθούν του θέματος αυτού οι αρμόδιες αρχές. Εδώ μιλάμε για δικήματα. Ε, είμαστε δημόσιοι λειτουργοί, ε, πρέπει να καταγγείλουμε αυτά τα δικήματα, αυτά τα εγκλήματα. Εγώ θα παρουσιαστώ σε κάποια εισαγγελία της Ιταλίας με αυτή την έκθεση. Ούτως ώστε κάποια εισαγγελική αρχή να επιληφθεί του θέματος. Γιατί είναι απαράλογο τέτοια εγκλήματα. Δεν θα μπορώ να πάω και στο ποινικό δικαστήριο πούμε, της Χάγης. Δεν μπορούμε τέτοια δικήματα να αφήσουμε ατιμόρυτα. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι μια κλασική κοινοβουλευτική συζήτηση αυτή. Και τώρα η κυρία Αντιτσέβιτς, η οποία για πρώτη φορά παίρνει το λόγο εδώ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, είναι ένα νέο μέλος, ε, παρατηρήτρια από την κουρατική αντιπροσωπεία. Σας καλωσορίσουμε και σας δίνουμε το λόγο. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πάντα δύσκολο να πούμε την αλήθεια. Τους αφήσαμε να πεθάνουν αυτούς τους ανθρώπους, παρά τα σήματα κινδύνου και εκτακτού ανάγκης, παρά το γεγονός ότι είχαν εντοπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή, δεν έγινε καν απόπειρα διάσωσης. Όλοι, εκτός από εννέα, αφέθηκαν να αποβιώσουν από πείνα, από τη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων και δύο μωρών. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να λέμε, αλλά αν παράλληλα αφήνουμε τον κόσμο να πεθαίνει, αυτό καταδεικνύει τη ματαιότητα όλων των μέτρων και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε σημαντικά. Αυτοί που φεύγουν από τη Λιβύη προφανώς δεν θεωρούνται προτεραιότητα, ούτε και η ευθύνη της ευρωπαϊκής δύναμης ή της δύναμης του ΝΑΤΟ. Να σημειώσουμε ότι δεν πρόκειται για μόνο με ένα περιστατικό. Ο ΙΕ υπολογίζει ότι τουλάχιστον 1.500 άτομα έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο το 2011. Και φαίνεται ότι ο κόσμος που ε, κάνει τέτοιες απελπισμένες κινήσεις για να φτάσει στην Ευρώπη, στη Δύση, θεωρούνται ότι είναι απειλή, ότι αποτελούν απειλή και όχι ότι έχουμε την ευθύνη να τους προστατεύσουμε να σας τονίσω ότι πριν από κάποια χρόνια στην Ιταλία ένας ε, ψαράς είπε στους δικαστές όταν είχε διασώσει κάποια άτομα ότι ποτέ δεν είμαι πιο βέβαιος ότι έκανα κάτι σωστό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βαπεντάη, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στρέικ για την έκθεσή της η οποία είναι πάρα πολύ σαφής και την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Είναι πραγματικά ε, ανατριχιαστικό ότι τη σήμερα ημέρα βλέπουμε εκατοντάδες άτομα να χάνονται ως πρόσφυγες στη θάλασσα, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό. Να υποστηρίξω την άποψη του κυρίου Μπουσουτήλ ότι προφανώς σημαντικό είναι να εξεταστούν οι αιτίε και να δούμε ποιο στέει, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μην συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον ξανά. Και θα ήθελα να σκεφτούμε από την άποψη αυτή τις ε, προτάσεις για την Eurosur. Είδαμε προτάσεις για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συστήματος Παρακολούθησης και Εποπτείας των Συνόρων για να υπάρξουν ε, εθνικά κέντρα συντονισμό προκειμένου να παρακολουθούμε την κατάσταση στην Ευρώπη και να υπάρχει και ένα σωστό δίκτυο επικοινωνίας. Εγώ θα ήθελα να απευθύνω έκκληση για να επικεντρωθούμε σε αυτά που μπορούμε να πράξουμε μέσω της Eurosure για να διασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα και θα κάνουμε συγκεκριμένα θετικά βήματα προς τα εμπρός. Και θα ήθελα αυτή την οδόν να ακολουθήσουμε παρά να ξοδέψουμε χρόνο για να απευθύνουμε, να κατηγορήσουμε τους υπευθύνους. Ο κύριος Μπρόντς, ευχαριστώ. Ποιο θα πρέπει να κατηγορήσουμε όταν 72 άτομα ξεκίνησαν σε μια ε, επικίνδυνη θαλάσσια αποστολή σε μια μικρή βάρκα. Οι λεβικοί, οι λεβικές αρχές αν ε, έπρεπε να τους ε, εκδιώξουν, θα έπρεπε να το έχουν κάνει αυτό με άλλη οδό. Αλλά αυτοί οι ίδιοι ήταν αυτοί που μπήκαν στην ε, βάρκα για να μπουν και να έρθουν στην χώρα, τη γη της επαγγελίας, στην Ευρώπη. Κατά δεύτερον, τα διάφορα σκάφη, τα διάφορα ελικόπτερα κατηγορούνται και η αποτυχία τους είναι όντως επιλήψιμη, αλλά να θυμόμαστε ότι αυτό το έκαναν γιατί ήξεραν ότι αν τους είχαν σώσει θα ε, είχαν ευθύνης οι χώρες τους, όπως το βλέπουμε σε διάφορες αποφάσεις ε, του δικαστηρίου. Φυσικά κατηγορούνται για την ε, μεταφορά τους στην Ευρώπη και η ευθύνη φυσικά βαραίνει και οποιοδήποτε άνθρωπο υποφελείται από την απελπισία των φτωχών του κόσμου, αλλά πιο πολύ από όλα η ευθύνη βαρύνει και τις πολιτικές και δικαστικές αρχές στην Ευρώπη, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, που ε, ανταποδίδουν ε, στους οικονομικούς μετανάστες, ε, τους επιβραβεύουν με το να μην τους ε, επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Και έτσι τους δίνουν ένα κίνητρο να μπαίνουν σε τέτοια επικίνδυνα σκάφη. Αν όλοι αυτοί οι υπεύθυνοι ε, διορθώνονταν, θα είχαμε λιγότερους μετανάστες. Για κολλήνω ο τελευταίος. Όλοι προλαλήσαντες είπαν πόσο τραγικά ήταν αυτά τα συμβάντα συμβάντα που μας παρουσίασε εκλαφυρά η κυρία Στρέικ. Μιλήσαμε για διακίνηση ανθρωπίνων όντων ε, στα χέρια του οργανωμένου εγκλήματος. Θα πρέπει κυρίως να κινηθούμε εναντίον αυτών των ανθρώπων, να σταματήσει αυτή η εμπορία ανθρώπων. Επίσης μιλήσαμε για διασταυρούμενες ευθύνες. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιους βαραίνουν. Αλλά το θέμα είναι γνωστό. Εγώ είμαι σικελός, όπως το ξέρουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ακόμα και σήμερα από τη Λιβύη, από την ε, ε, Αίγυπτο έρχονται ε, τέτοιε βάρκες, τέτοια σκαφίδια και φτάνουν στη Λαμπεντούζα κτλ. Εμείς τους αποβιβάζουμε και μετά από 48 ώρες τους μεταφέρουμε αλλού. Εμείς πολλές φορές ε, κάναμε, θέσαμε αυτό το θέμα στην, ε, στην Ολομέλεια και στην τελευταία σύνοδο του Στρασβούργου. Ε, θέλουμε να δούμε πού βρίσκεται η ευθύνη. θέλουμε να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Κυρία Στρίκ, κύριε Σαντίνη, καταρχάς, βασικό θέμα είναι οι διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνοριακών όμορων χωρών. Ας πούμε με τη Λιβύη εντάξει δεν μπορούμε να έχουμε, αλλά μπορούμε να έχουμε την Τινησία. Ας πούμε με την Αίγυπτο. Θεωρούμε ότι μπορεί να είναι ένας αξιόπιστος συνομιλητής. Αν δεν λύσουμε αυτά τα θέματα των διμερών συμφωνιών, αποκλείεται να επιλύσουμε το πρόβλημα τη διακίνηση ανθρώπων. Θα αντιμετωπίζεται εδώ στην Ιταλία, στη Μάλτα, στην Ισπανία. Θα είναι ανεπίλητο πρόβλημα και αυτή η ευθύνη είναι σαφώ τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν δείχνει την αλληλεγγύη. Την αλληλεγγύη που όλοι θέλουμε τελευταίο σχόλιο, αν θέλετε να αντιδράσετε κυρία Στρίκ στα σχόλια που ακούσατε, στις ερωτήσεις που ακούσατε για την έκθεση. Κυρία Στρίκα, ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις στην παρουσίασή μου, για τις αντιδράσεις στην παρουσίασή μου, για τα συγχαρητήριά σας και μερικές φορές και για τις επικρίσεις σας. Αλλά από όλα μαθαίνουμε. Θέλω να τονίσω ήδη από την αρχή ότι αυτό που είπε ο κύριο Μπουσουτήλ είναι σωστό, ότι έκτοτε, μετά από αυτό το περιστατικό, δηλαδή έγιναν και άλλα ατυχήματα. Ε, άρχισα την παρουσίασή μου την προηγούμενη με αυτό. Πέρυσι, 1500 άτομα πέθαναν στη Μεσόγειο. Ο λόγος που κάνουμε αυτή την ε, ενδελεχή αξιολόγηση είναι γιατί θέλουμε να μάθουμε από αυτό το ατύχημα, ε, ώστε να αποφύγουμε τέτοια ατυχήματα στο μέλλον. Αλλά πρέπει παράλληλα να κινηθούμε ε, και πρέπει και να μάθουμε επακριβώ τι έγινε, ούτω ώστε να μπορέσουμε να μάθουμε. Επομένω, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα γεγονότα. Ποιο ήταν υπεύθυνο, γιατί δεν υπήρξε αποτελεσματική απόκριση, ενώ προφανώ ε, φύγανε σήματα κινδύνου. Και μετά, αφού λύσουμε τα πρώτα θέματα αυτά που σα ανέφερα, μπορούμε να δούμε τι συστάσει μπορούμε να κάνουμε με συμφωνία με τα κράτη-μέλη ή, εν πάση περιπτώσει, με τις διεθνείς οργανώσεις, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον θα υπάρξει αποτελεσματική απάντηση. Επομένως, ψάχνουμε τι έγινε στο παρελθόν, τόσο ώστε να αποφύγουμε αντίστοιχα πράγματα στο μέλλον. Ο κ. Μπουσουτήλ είπε ότι οι διακινητές είναι οι ένοχοι. Προφανώς είναι οι ένοχοι. Αλλά συμφωνώ και με την κυρία Σαρτζεντίνη ότι πρέπει να κοιτάξουμε και πάρα πέρα, πέρα από τους διακινητές. Γιατί οι διακινητές ε, χρησιμοποιούν αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβη, στον Καντάφη και στους ε, αντάρτες. Και είναι, ας πούμε, ε, άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τον εμφύλιο στην ε, Λιβύη. Άλλοι πολίτες ε, μπόρεσαν να φύγουν από τη Λιβύη. Ε, αυτοί δεν μπόρεσαν οι συγκεκριμένοι. Επομένως, πρέπει να ψάξουμε όλους τους παράγοντες, όλες τις αιτίες που συνέβαλαν τόσο ώστε να συμβεί αυτό το γεγονός και αυτοί οι απελπισμένοι άνθρωποι να πάρουν την απόφαση να ξεκινήσουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι στη θάλασσα και να βρεθούν σε αυτήν την κατάσταση απελπισίας και εγκατάλειψης από τους άλλους. Αυτό που συμβαίνει ε, και στην ανοιχτή θάλασσα είναι και ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δεν είναι κάτι εξοεδαφικό, κάτι που δεν μας αφορά, που δεν είναι αρμοδιότητά μας. Είμαστε και εμείς και τα επιμέρους κράτη-μέλη συνυπεύθυνα. Τώρα έχουμε κοινά σύνορα ε, και επομένως πρέπει να ψάξουμε να βρούμε κοινέ λύσεις σε αυτά τα προβλήματα. Θέλω λοιπόν να ζητήσω και να κάνω έκκληση ακόμα μια φορά, ούτω ώστε να υπάρξει ένα δεσμευτικό πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε και άλλα θέματα βεβαίω, αλλά ας ξεκινήσουμε αυτό το πρωτόκολλο ε, για τη Μεσόγειο και μετά μπορούμε να το επεκτείνουμε, ας πούμε, στον, σε άλλες περιοχές. Έχουμε και τις άλλες περιοχές υπόψη. Αλλά δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε χωριστά τα επιμέρους προβλήματα. Θέλουμε να ξεκινήσουμε απλώς την προσπάθεια. Ε, μιλάμε για την ποινικοποίηση αυτών των ανθρώπων, ε, των διακινητών ας πούμε. Αλλά έχουμε δει ας πούμε εμπορικά σκάφη τα, οποία διασώζουν απελπισμένους και τα οποία αντιμετωπίζουν κυρώσεις. Γιατί τους υποψιαστήκαμε ότι ε, μπλέκονται σε διαδικασίες λαθρεμπορίου και διακίνησης ανθρώπων. Παίζουν τόσα πολλά πράγματα ρόλο ούτως ώστε και τα εμπορικά σκάφη και τα ψαράδικα να διστάζουν να δώσουν συνέχεια και να ανταποκριθούν στα σήματα κινδύνου. Όλα αυτά πρέπει να τα συνεκτιμήσουμε. Και επίση πρέπει να δείξουμε στα κράτη που είναι στην πρώτη γραμμή του πυρό ότι δεν είναι μόνα του. Από τη στιγμή που αυτά κάνουν κάτι για να διασώσουν τέτοιου ανθρώπου, ε, τους λέμε ότι συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις ε, και ότι μετά όμως δεν θα αναλάβουν μόνοι τους την ευθύνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εσείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχετε την ε, δυνατότητα να ξεκινήσετε αυτή την έρευνα για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρωτόκολλο και πώς μπορούν να ξεκαθαριστούν οι κοινέ ευθύνε. Αναφέρθηκε το Eurosur ως η λύση. Και εγώ έχω πολλές προσδοκίες από μια τέτοια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Φυσικά εξαρτάται και από το τι κάνουμε με αυτές τις πληροφορίες. Αν μπορούμε να ανοιχνεύουμε πολύ μικρά σκάφη, ε, μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να έχουμε και μια σωστή συνέχεια με βάση το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο και να μην χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να επαναπροωθούμε αυτούς τους ανθρώπους ή για να αποποιούμαστε τις ε, ευθύνες και να τις ε, ρίχνουμε στα βορειοαφρικανικά κράτη. Ε, θέλουμε να υπογράψουμε συμφωνία με, τις, με αυτές τις χώρες και να τους πούμε ε, κρατήστε αυτούς τους μετανάστες εκεί. Αλλά μπορεί τα ανθρώπινα τους δικαιώματα να παραβιάζονται. Ε, μην ξεχνάμε ότι ποια είναι η αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο για να εξασφαλίσει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ελπίζω να συνεργαστούμε και στο μέλλον για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ για την ανταλλαγή απόψεων. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι ένα θέμα ανησυχίας για όλους μας, για, για όλους εμάς που εκπροσωπούμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεργαστούμε με τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Κύριε Σαντίν, ένα τελευταίο, μια τελευταία κουβέντα θέλετε να πείτε. Ένα λεπτό, Πρόεδρε. Να τονίσω και εγώ αυτά που είπε η κυρία Στρίκ, ότι το πρόβλημα μπορεί να απασχολεί καταρχήν λίγε χώρε τη Μεσογείου. Αλλά παρόλα αυτά είναι ένα πρόβλημα όλων μα. Γιατί, Γιατί καταρχά είναι ηθικό το πρόβλημα, ηθικό το θέμα. Όταν πεθαίνουν άνθρωποι, νομίζω ότι κανένα κρατό μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή του Συμβουλίου τη Ευρώπη τέλο πάντων δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν το αφορά αυτό το θέμα και δεν έχει καμία ευθύνη. Δεύτερο, για πρακτικού λόγου. Ε, Όντω, αποβιβάζονται στην Ιταλία και στην Ισπανία αυτοί οι άνθρωποι καταρχήν. Αλλά το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των λαθρομεταναστών θέλουν συνεχεία να πάνε σε άλλε χώρε, στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Σουηδία. Βοηθήστε μα λοιπόν να ελέγξουμε το φαινόμενο για πρακτικού λόγου και για το συμφέρον όλων μα. Πώ μπορούμε να συνεργαστούμε. Ε, εδώ δεν ήρθαμε μπροστά σα για να ξεκινήσουμε μια πολεμική και για να ξεφορτώσουμε ευθύνε. Ε, θέλουμε απλώ να συνεργαστούμε. Εμεί κάνουμε ό,τι μπορούμε από πλευρά Συμβουλίου τη Ευρώπη. Εμεί έχουμε όμω περιορισμένε οικονομικέ δυνατότητε, για να μην σα πω καμία. Εμεί ασχολούμαστε με ανθρώπινα δικαιώματα και απλώ ε, ε, απευθυνόμαστε στι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών. Εσεί όμω έχετε πόρου ε, για να παρέμβετε. Εσεί είσαστε διαιτητή εκεί. Μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένε παρεμβάσει και γίνονται συγκεκριμένε παρεμβάσει αν υπάρχουν πόροι. Μια τελευταία σύσταση που αφορά όλου. Α ξανανοίξουμε το θέμα των ασύλων και των πολιτικών για το άσυλο, λαμβάνοντα υπόψη ότι οι αιτούντε σε άσυλο δεν είναι αυτοί που φτάνουν ένα-ένα. Μερικέ φορέ ε, φτάνουν 300-400 μαζί. Μαζικά. Ε, τέλος, οι διμερεί συμφωνίε που εσεί εγκρίνετε στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Διμερεί ε, συμφωνίε σημαίνει συμφωνία μεταξύ μιας ε, χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας τρίτης χώρας, έτσι. Ε, υπήρξε μια αρνητική συμφωνία που οδήγησε και σε μια απόφαση του δικαστηρίου ανθρωπινών δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να σπρώξουμε πίσω στη θάλασσα κανέναν. Δεν μπορούμε να διώξουμε κανέναν. Αυτά και ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους μας, την κυρία Στρίκ, τον κύριο Σαντίνη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ και προσβλέπουμε στη συνέχιση της συνεργασίας μας. And no further delay, we proceed to the following point. Μπορούμε να περάσουμε χωρίς καθυστέρηση στην επόμενη έκθεση, η οποία ουσιαστικά αφορά την ε, παρουσίαση της, Επιτροπή, της Αντιπροσωπείας Επιτροπής Λίμπες στην Ουάσιγκτον 18 έως 22 Μαρτίου. στόχος ήταν πρώτα απ' όλα να ε, δουν ε, τις πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Δεύτερον, την υλοποίηση των συμφωνιών ε, αμοιβαίας νομικής συνδρομής και έκδοσης και το TFTP. Τρίτο θέμα ήταν απειλές στην ελευθερία έκφρασης, ελευθερία χρήση του διαδικτύου αλλά και προστασία της ιδιωτικής σφαίρας στο PNR. Τα στοιχεία δεδομένων επιβατών ήταν και αυτό ένα θέμα συζήτησης. Θα μας πει τα σχετικά ο εισηγητής μας ο κ. Άλβαρο και μετά θα ξεκινήσει για μισή ώρα μισή ώρα συζήτηση. Κύριε Άλβαρο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εξ όσων κατάλαβα, η έκθεση δεν έχει διανεμηθεί ακόμη. Ο Πρόεδρος. Ναι, μου είπαν ότι θα διανεμηθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ τις επόμενες ημέρες. Μάλιστα, λέει ο κύριος Άλβαρο. Θα την έχετε σύντομα, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει στην ημερήσια διάταξη ε, θα ήθελα εν συντομία να παρουσιάσω αυτά που πράξαμε. Καταρχάς, ε, να σας πω ότι η σύνθεση της αντιπροσωπείας ε, περιλάμβανε εμένα, την Βαρόνι Λάντφορτ, τον κύριο Σόνικ, τον κύριο Τρούτσα, την κυρία Ρομέρο Λόπες, τον κύριο Δίας Δεμέρα, Κισίπερ, Μέλο, Παπα-Νικολάου, Άλμπρεχτ και ασφαλώς την Κλέρ Βέλς που είναι επικεφαλής του γραφείου μας στην Ουάσιγκτον. Ατουάν Καουίν, Ελίνα, Πέτρα Γκέτς. Θα ήθελα λοιπόν εξ αρχής να τους ευχαριστήσω για την υποστήριξή τους, για τη δουλειά που έκαναν στην Ουάσιγκτον. απέδειξαν πόσο ικανή είναι η βοήθεια της γραμματείας και πόσο αποτελεσματική είναι η γραμματεία. Θα θυμάστε ποιοι είναι οι στόχοι της αντιπροσωπείας. Συμμετείχαμε σε μία διάσκεψη για την ιδιωτική σφαίρα και την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων στις 19 Μαρτίου. Τέσσερα μέλη της ΛΥΜΠΕ συμμετείχαν ως ομιλητές και ο σκοπός ε, της αντιπροσωπείας ήταν να γίνει μια συζήτηση βάθος με τους ε, Αμερικανούς ομολόγους ε, για τις πρόσφατες εξελίξεις μετά από την διάσκεψη της 19 Μαρτίου, εφαρμογή της κοινή συμφωνίας και των συμφωνιών έκδοσης και σε ό,τι αφορά θέματα ελευθερίας έκφρασης και τέλος η συμφωνία για τα νόματα των επιβατών αποτέλεσε ένα θέμα το οποίο συζητήθηκε από την αντιπροσωπεία. Στο μεταξύ έχει ψηφιστεί ε, οι συναντήσεις τώρα με το Υπουργείο Οικονομικών, Εσωτερικών, Εμπορίου, Δικαιοσύνης και θεωρώ ότι στο Λευκό Οίκο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντηση με τον κύριο Μπραντον, που είναι υπεύθυνο για θέματα ασφάλεια, τον Ντάνιελ Βάιτς, επικεφαλής για την πολιτική για το διαδίκτυο και αυτός ε, ε, συστήνει στον πρόεδρο Ομπάμπα πώς να προχωρήσει με τη σχετική πολιτική με την Επιτροπή Ομοσπονδιακού Εμπορίου. Συζητήθηκε θέματα με το Κέντρο της Δημοκρατίας, με το Ευρωπαϊκό Σχετικό Ινστιτούτο και νομίζω ότι συμπερασματικά ως follow-up μπορούμε να πούμε ότι οι συναντήσεις ε, της αντιπροσωπείας αποτέλεσαν μια πρώτη αντίδραση για το μακέτο μεταρρύθμισης για τα προσωπικά δικαιώματα και για την λευκή ε, βίβλο της Ουάσιγκτον. Και όλα αυτά μας έδωσαν ε, μια ιδέα για το πώς μπορούμε να συντονιστούμε. Οι συναντήσεις επίσης αποτέλεσαν μία πλατφόρμα για τις ε, αμερικανικές πρακτικές. Ε, συναντήθηκαν κάποιοι συνάδελφοι με προσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ασφαλώς την προσωπία κατάφερε να συζητήσει περαιτέρω την ε, συμφωνία PNR και τη USTFP και τις συμφωνίες για την προστασία των δεδομένων. Επίσης πρόσφεραν να φόρουμ για να εκφραστούν στους Αμερικανούς οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου για κάποια σημεία των συμφωνιών. Εκτίμηση λοιπόν ε, της ε, συμφωνίας TFEP μπορεί να ε, δούμε τα σχετικά συμπεράσματα. Ξέρω ότι προγραμματίζεται για μέσα Ιουνίου να τα συζητήσουμε, αλλά για να... Να σας πω ότι υπενθυμήθηκε ότι θα πρέπει να συνεχίσει ο διατλαντικός ε, διάλογος για θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ε, επίσης σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και θέματα ιδιωτικής σφαίρας. Αυτό που καταφέραμε να συμφωνήσουμε και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ νέου για την πρωτοβουλία και της γραμματείας που μας συνόδευε. Αυτό λοιπόν που πετύχαμε είναι να εγκαθιδρύσουμε να βεβαιωθούμε ότι πρόκειται για την πρώτη πολλών συναντήσεων, όχι για μια μεμονωμένη συνάντηση και ενδεχομένως να γίνει ακρόαση στο φθινόπωρο του 2012 στις ε, Βρυξέλλες και μια σχετική εκδήλωση του 2013 την Άνοιξη στην Ουάσιγκτον. Συνολικά πρέπει να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα αντιμετωπίσαμε και κάποιες δυσκολίες, ε, βρήκαμε κάποιους κοινού τόπους και νομίζω ότι είπα κατανοούν καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη της Επιτροπής μας είναι αυτοί που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για περαιτέρω συναντήσεις, συζητήσεις και για τη συνεργασία μεταξύ των ΙΠΑ και της Ευρώπης στους ε, προκαθορισμένους τομείς. Αν έχετε ερωτήσεις, βλέπω ότι είναι εδώ και κάποιοι συναδελφοί που μου συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία. Ίσως και αυτοί θέλουν κάτι να προσθέσουν, να με διορθώσουν σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Σας ευχαριστώ κύριε Άλβαρο, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ας κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Κάποια μέλη της αντιπροσωπείας που συμμετείχαν στην αποστολή στην Ουάσιγκτον έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Δίας Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενα του κυρίου Άλβαρο. Τα είπε πάρα πολύ συνοπτικά και συνθετικά. Πράγματι μου και εγώ στην αντιπροσωπεία. Ήταν μία ακόμη από τις αντιπροσωπείες στις οποίες συμμετείχα και ήταν μία ακόμη ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα ζητήματα όπως ε, είναι η Συμφωνία PNR, η προστασία των ε, δεδομένων, της θετικής σφαίρας ε, και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι για τις μελλοντικέ συναντήσεις και αντιπροσωπείες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα ζητήματα. Λίγο, πολύ λίγο ενδιαφέρον είδαμε να δείχνουν οι βουλευτές. Οι βουλευτές φαίνεται ότι οι δικές μας απόψεις δεν τους ενδιαφέρουν και ιδιαίτερα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον, γιατί είναι καλό να συνεννοούμαστε με τους ομολόγους μας και όχι με εκπροσώπους κάποιων κυβερνητικών οργανισμών. Στο Υπουργείο Οικονομικών, ε, στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, Ασφάλειας, Άμυνας, στο Λευκό Οίκο ε, και με το Ομοσπονδιακό Τμήμα Εμπορίου. Είχαμε επαφές, είχαμε κάποια συνεννόηση. Νομίζω ότι και η συνάντησή μας στο φθινόπωρο θα είναι πάρα πολύ θετική, ένα ακόμη βήμα προσέγγισης. Αυτό που δεν ξέρω αν σχολείς ο κύριος Άλβαρο είναι ότι η πρόοδος για την αμερικανική πλευρά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσουν από μια νομοθετική μεταρρύθμιση δεν θέλουν νομοθετική μεταρρύθμιση. Για θέματα που όμως εμάς τόσο πολύ μας ενδιαφέρουν. Ελπίζω πάντως να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε τις σχέσεις της Δημερής. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να επιβεβαιώσω όλα αυτά τα οποία είπε ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας ε, στην ε, Ουάσιγκτον. Διότι πράγματι το ενδιαφέρον των Αμερικανικών αρχών ήταν ε, πάρα πολύ καλό, πολύ μεγάλο. Ήθελα να πίσω όλα τα αιτήματα της αντιπροσωπείας μας, αλλά πράγματι σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση ε, της συμφωνίας, γιατί είμαστε ένα από τα συμβαλόμενα μέρη, Εκεί πράγματι ε, θέλω να πω ότι δεν ήταν απλά ομολογή μας ε, οι Αμερικανοί. Ένα τέτοιο θέμα είναι ένα θέμα που ε, βρίσκεται και στην ε, έδρα του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Στην προηγούμενη επίσκεψη, όχι αυτή, η προηγούμενη ήταν πολύ χρήσιμη, γιατί στο μεταξύ παρουσίασε ο κύριος Ομπάμα με έκθεση για την προστασία των δεδομένων, άλλαξε έτσι η ευαισθησία σε σχέση με αυτά τα θέματα, αλλά δεν είχαμε με τους ε, Αμερικανούς ε, βουλευτές του Κογκρέσου επαφή. Δεν ξέρω αν εμείς εδώ θα μπορούσαμε να καλέσουμε μέλη του Κογκρέσου, εδώ, στο Κοινοβούλιο, και συγκεκριμένα μιλώ για τους ε, βουλευτές που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα της προστασίας των δεδομένων, γιατί υπήρχαν πολύ συγκεκριμένα θέματα τα οποία αυτή τη στιγμή συζητούνται στο Κογκρέσο και εμεί δεν είχαμε τη δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή με αυτού του ανθρώπου και να τα συζητήσουμε όταν πήγαμε εκεί. Κάθε φορά που πηγαίνουμε στη ΣΥΠΑ, δεν είναι φυσιολογικό στο Κογκρέσο τον ΗΠΑ να εμφανίζεται μια πλήρης αντιπροσωπεία τη επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Γι' αυτό το φυσιολογικό είναι ένας, ένα μέλο του Κογκρέσου με ένα μέλος ε, του Κογκρέσου. Δεν πάει μια ολόκληρη επιτροπή με, για να δει ε, ένα μέλο του ε, Κογκρέσου. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να βελτιώσουμε κάπως τα πράγματα, να βελτιώσουμε και τι γνώσει μα, να έρθουμε σε επαφή δηλαδή με μέλη του Κογκρέσου για να συνεχίσουμε αυτή την πρόοδο, γιατί πράγματι θα υπάρξει αλλαγή τη νομοθεσία στο μέλλον, ίσως και από τι δύο πλευρέ. Για αυτού τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι ε, μεταξύ άλλων και τα δικαιώματα των καταναλωτών, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά στην, ε, στον τρόπο με τον οποίο κάποια πράγματα. Πανικολάου. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον επικεφαλής ε, κύριο Άλβαρο για την πρωτοβουλία του, τη γραμματεία, όλους όσοι συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία αυτή. Όντως ήταν η δεύτερη φορά που συμμετείχα σε μια τέτοια αντιπροσωπεία και όντω. και εγώ αισθάνθηκα και αυτό το προσθέτω σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι ότι προσεγγίζουμε. Παρά το γεγονός ότι είπα έχουν διαφορετική προσέγγιση σε πολλά ζητήματα σε σχέση με τη δική μας προσέγγιση. Πριν από 10 χρόνια η επίθεση της ΕΝΑ Σεπτεμβρίου, της 11 Σεπτεμβρίου αποτέλεσε ένα σημαντικό παράγοντα για την αλλαγή της στάσης ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων κτλ. Όλοι τα γνωρίζουμε αυτά. Παρά όλα αυτά, ε, όντως προσεγγίζουν οι απόψεις μας, συγκλίνουν οι απόψεις μας και φυσικά πολλά ακόμα παραμένουν να συζητηθούν. Ήταν καρποφόρες στις συζητήσεις μας, ήταν πολύ καλές πολλές νέες επαφές που κάναμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καλέσαμε και κάποιους να έρθουν εδώ για να συντηρηθούν αυτές οι καλές επαφές στο εγγύς μέλλον. Ε, όχι μόνο σε αμερικανικό αλλά και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μέλλον να προσπαθήσουμε και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Διαθεμέρα και η κυρία Λόπες. Είναι σημαντικό να γίνονται καλύτερες συζητήσεις σε πολιτικό όμως επίπεδο. Σε όλες μας τις συναντήσεις ε, μας έλεγαν ότι ναι, συμφωνούμε, καταλαβαίνουμε τι λέτε, γνωρίζουμε τα τεχνικά ζητήματα, αλλά είναι πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν και αυτό θα πρέπει να το συζητήσετε με τους ε, υπευθύνους του Κογκρέσου και με τους συναδέλφους σας. Άρα, για το μέλλον, και εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθούν, να συνεχιστούν αυτές οι αντιπροσωπείες, να έχουμε την στενότερη δυνατή επαφή, να προσπαθήσουμε να υπάρξουν πολιτικές συμφωνίες στην επόμενη συνάντησή μας και στη ΣΥΠΑ, αλλά και εδώ σε ενδεχόμενη ακρόαση και σε άλλες συναντήσεις. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Σας ευχαριστώ. Εγώ δεν είμαι και τόσο αισιόδοξη όπως οι υπόλοιποι συνάδελφοι σε ό,τι αφορά το θέμα. Σε ό,τι αφορά την προσέγγιση για τα προσωπικά δεδομένα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Θα θέλαμε να σας ε, πούμε ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτό έχει φτάσει σε όλες τις ε, κλίμακες της ε, κυβέρνησης και ότι δεν θα υπάρξει ενιαία σχετική ε, νομοθεσία στις ΕΠΑ για την προστασία των δεδομένων. Θα δούμε λοιπόν τελικά ποιος θα επικρατήσει. Και αυτό που με ενοχλεί είναι το εξή στη συζήτηση με τη ΕΠΑ, η οποία ασφαλώς και είναι απαραίτητη. Αν μας διευκρινίζουν ότι ε, υπάρχει κάποια άποψη, γιατί τελικά ε, με ποιους θα πρέπει να μιλήσουμε, με την κοινωνία των πολιτών, με τους πολιτικούς. Καλό θα ήταν ε, να μην είχαν μόνο κάποιες ομάδες, κάποια κόμματα, μία άποψη. Καλό θα ήταν ως κοινοβούλιο να είχαμε μία ενιαία θέση, αλλά κοιτάξτε, βρισκόμαστε την αρχή της συζήτησης. Συνολικά θα πρέπει να ξεκαθαρίζουμε, για παράδειγμα, να πω ότι υποστηρίζω την κυρία Ρέντινγκ που τόνισε ότι πρόκειται για μια βασική αξία την οποία θα πρέπει να προσπίσουμε και όχι για μια λεπτομέρεια και ότι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κοιτάξουμε πόσο σημαντική είναι η προστασία των δεδομένων, πόσο σημαντικά είναι τα οικονομικά συμφέροντα, θα πρέπει να βρούμε μια ισορροπία και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο εξωτερικό και θα πρέπει να κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσει με τους εταίρους μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Herbert. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αλεξάνδρα Άλβαρο, τον επικεφαλιστή της προσωπίας ο οποίο ε, τα συνόψισε όλα πολύ αποτελεσματικά. Μία προστίκη, επιτρέψτε μου, Εν συντομία, η διάσκεψη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μάλλον η διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προστασία των δεδομένων για τις σχετικέ μεταρρυθμίσεις ε, σε αμφότερε πλευρές ε, του Ατλαντικού και σε σχέση με την ε, συνεργασία που χρειάζεται μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού είναι πολύ σημαντικό σημείο και το σημείο που έθιξε ο κύριος Αντιευθεμέρα και άλλοι, ότι αυτή η ενίσχυση της θεματικής συνεργασίας είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βρει συνέχεια. Το τονίζω αυτό. Και ως εκ τούτου, μετά από την αντιπροσωπεία, την αποστολή αυτή, είδαμε ότι στην ακρόαση για το πακέτο προστασίας των δεδομένων, το οποίο θα συζητήσουμε το αύριο, στην ακρόαση τον Οκτώβριο θα καλέσουμε και εκπροσώπους από τη ΣΥΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να γίνει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε εκπροσώπους, να καλέσουμε εκπροσώπους από τη ΣΥΠΑ και από το Κογκρέσο για να μιλήσουμε για τα ελάχιστα πρότυπα σε ό,τι την προστασία των δεδομένων και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και ως εισηγητής του κανανισμού που θα συζητήσουμε αύριο. Είναι σημαντικό τώρα να γίνει ένας διατλαντικός διάλογος. Μέσω μιας προσέγγισης των προτύπων και πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα äh, da angeht, ähm, Ότι στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδο και τα μηνύματα είναι θετικά. Σε ό,τι αφορά και την αστυνομική συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνη, πρέπει να σα πω ότι είμαι κάπως απεσιόδοξος είμαι. Ασχολούμαι με τέτοια θύματα και θα πρέπει να σας το πω, το λένε και άλλοι συνάδελφοι νομίζω, ότι το feedback που λαμβάνουμε από τις διαπραγματεύσει δεν ε, μας δίνει λόγους αισιοδοξία για την προσέγγιση σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά πρότυπα. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουμε πετύχει σε καμία περίπτωση το στόχο μας. Δεν θα έχουμε πετύχει αυτό που θα θέλαμε να έχουμε πετύχει. Θα πρέπει λοιπόν μεταξύ βουλευτών να γίνεται συχνότερη ανταλλαγή απόψεων και θα πρέπει να σκεφτούμε και νέους τρόπους επικοινωνίας, όχι μία φορά το χρόνο να πηγαίνουμε στην Ουάσιγκτον και να συναντιόμαστε για μία ώρα με τον ε, αντίστοιχο ομόλογο μας ε, ίσως βιντεοδιασκέψεις να διοργανώνονται, να τους προσκαλούμε εδώ στις Βρυξέλλες. Όλα αυτά να τα συζητήσουμε πιο πολύ για να έχουμε πιο άμεση επαφή με τους εκπροσώπους από την Ουάσιγκτον. Και τώρα δίνουμε το λόγο στον κύριο Άλβαρο. Δεν βλέπω να θέλει κανένας άλλος το λόγο. Αν δεν θέλει κανένα να μιλήσει, να σας πω ότι έχουμε προβλέψει στις αρχές του φθινοπόρου, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διαποθές, διακοπές, να κάνουμε μία από αυτές τις κλασικές συναντήσεις ανάμεσα στα μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωκοινοβουλίου, ούτω ώστε να δούμε πώς αναπτύσσεται ο χώρος της δικαιοσύνης, ελευθερίας και εσωτερικών υποθέσεων. Ε, προβλέπεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Μέχρι στιγμής έχουμε συγκεντρώσει κάποιες εμπειρίες. Θέλουμε να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Προβλέψαμε λοιπόν επευκαιρία αυτή τη συνάντηση ε, του Σεπτεμβρίου να καλέσουμε και μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου για να συμμετάσχουν και της Αμερικανικής Κυβέρνησης για να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση, ούτως ώστε αυτή η αρχή που έχουμε θεσπίσει, ότι θα πρέπει όλο και περισσότερο αυτός ο κοινοβουλευτικός διάλογος μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων αλλά και του Αμερικανικού Κογκρέσου να γίνεται όλο και καλύτερος. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί περιοδικά. Θα τους αποστείλουμε πρόσκληση. Το λέμε από τώρα. Κύριε Άλβαρο, για να κλείσετε αυτή την ενημέρωση, σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε, μπορώ να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ για την ε, επικοδομητική σας δουλειά όσους συμμετείχατε στη Washington. Θέλω, έχω ήδη, έχω ήδη εκφράσει την ε, ευγνωμοσύνη μου στα μέλη της ε, γραμματείας. Για τους Αμερικανούς ομολόγους μας, άντρες και γυναίκες, καλή ιδέα να τους προσκαλέσουμε. Νομίζω ότι θα πρέπει να τους δείχνουμε ότι δεν μας απογοητεύει το γεγονός ότι δεν παρίστανται στη συνεδρία όταν ήμασταν στη Ουάσιγκτον. Μην ξεχνάτε όταν τους προσκαλέσετε ότι τον Νοέμβριο έχουμε τις εκλογές στην Αμερική. Ίσως λοιπόν να είναι λίγο απασχολημένοι. Έχω αυτό το θέμα ας που θα ήθελα να σας πω. Εναλλακτικά θα μπορούσατε να προσκαλέσετε τους ανώτατους ε, υπαλλήλου, γιατί στο νομοθετικό αμερικάνικο σύστημα μάθαμε από τις επαφές μας τα τελευταία χρόνια ότι οι ανώτατοι υπάλληλοι εμπλέκονται εκ του και στην νομοθετική διαδικασία και οι, τα μέλη του Κογκρέσου ε, βασίζονται σε αυτούς στο Κογκρέσο, όπως θα μπορούσαμε, όπως και εμείς εδώ ας πούμε. Επομένως, η νομοθεσία ε, κινείται συχνά από τέτοιους ανώτατους αξιωματούχους. Ως λύση, ας πούμε, δεύτερη, ως λύση καταφυγής, α, αν δεν έρθουν, ας πούμε, τα μέλη του Κογκρέσου, ε, να μπορέσουν να έρθουν ανταυτόν οι ανώτεροι υπάλληλοι. Δεν θα πρέπει εμείς να είμαστε απρόθυμοι να συναντηθούμε με αυτούς, γιατί και αυτοί συμμετέχουν στην νομοθετική διαδικασία. Ε, σκοπός μας είναι να υπάρξει διάλογος. Ας μπορέσουμε, ας μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε λοιπόν. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αμερική θα λάβουν χώρα εκλογές ε, το φθινόπωρο. Δεν θα το ξεχνάμε, δεν θα το ξεχάσουμε όταν ε, ετοιμάσουμε τις, προσκλήσει. προσκλήσεις. Αυτά προς το παρόν. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σε έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που έχει δοθεί στον Κυριάκο Τριανταφυλλίδη για την ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα του ασύλου. Είναι μια πρόταση της Κομισιόν στον τομέα του ασύλου για τον καλύτερο επιμερισμό της ευθύνης, περισσότερη αμοιβαία εμπιστοσύνη, υιοθετήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 η πρόταση της Κομισιόν, το Συμβούλιο έφτασε στα συμπεράσματα για ένα κοινό πλαίσιο για μια πραγματική και πρακτική αλληλεγγύη απέναντι στα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες πιέσεις ε, στο δικό του σύστημα ασύλου, ε, που συμπεριλαμβάνουν και μικτές μεταναστευτικές ροές. Το Μάρτιο του 2012. Έχουμε λοιπόν αυτή την έκθεση της ιδίας πρωτοβουλίας για τον κύριο Τριανταφυλλίδη που απεικονίζει την αντίδραση του Κοινοβουλίου στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Θα ακούσουμε τον κύριο Τρενταφυλλίδη και συνεχεία θα ξεκινήσει μια συζήτηση. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και ένα άλλο σημείο στη Μέσια Διάταξη για το συντονιστή κατά της τρομοκρατίας, τον κύριο Ζιλ Κερκόφ, ο οποίος θα έρθει σε λίγο. Μην ξεχνάτε λοιπόν ότι έχουμε και αυτό το σημείο στη Μέσια Διάταξη θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το θέμα του κυρίου Τριανταφυλλίδη και το θέμα του κυρίου Ντεκερκόφ, ούτως ώστε αμέσω μετά να αρχίσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Κύριε Τριανταφυλλίδη. Γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσει για τη διαμόρφωση ενός κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου μας απασχολούν χρόνια τώρα και οι διαφορές μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν είναι πάντα εύκολο να γεφυρωθούν. Πρόθεση μου μέσω αυτής της έκθεσης δεν είναι να προσθεθεί επιπλέον πολυπλοκότητα και ασάφεια σε αυτή τη διαδικασία, αλλά του αντίον ελπίζω να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πραγματικού χώρου προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών. Αυτά δεν είναι αφηρημένες έννοιες οι οποίες αρκεί να αναφέρονται μεν ρητά αλλά να εγκαταλείπονται έπειτα στην πράξη όπως έχουμε δυστυχώς συχνά διαπιστώσει. Αντιθέτως, η αλληλεγγύη και η δίκαιη κατανομή των ευθυνών είναι αρχές που κατοχυρώνονται στο άρθρο 80 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ορίζει ότι οι πολιτικές της Ένωσης που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο και η εφαρμογή τους διέπονται από την αρχή της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων και στο οικονομικό επίπεδο. Όποτε απαιτείται, οι πράξεις της Ένωσης που θεσπίζονται βάσει του παρόντος κεφαλαίου περιέχουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της εν λόγω αρχής. Δεδομένου ότι η ερμηνεία αυτών των αρχών μπορεί να διαφέρει και διαφέρει από όσο έχει διαφανεί μέχρι σήμερα, είναι σημαντικό να δουλέψουμε για να απαντήσουμε στο τι σημαίνει αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή ευθυνών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσουμε ένα έμπρακτο και αποτελεσματικό μηχανισμό και να μην καθίστανται οι έννοιες αυτές κενές νοήματος πια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να επισημανθεί πως αλληλεγγύη και κατανομή ευθυνών δεν σημαίνουν μετατόπιση ευθυνών. Δεν τίθεται ζήτημα απαλλαγή των κρατών μελών από τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και το ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το άσυλο. Αυτό που έχει σημασία εν προκειμένου είναι να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο δίκαιης κατανομής ευθυνών που θα εξοπλίσει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου με συγκεκριμένα μέσα και διαδικασίες με στόχο τη στήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δυσανάλογες πιέσεις και υψηλές δαπάνες στον τομέα του ασύλου, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης ή της δημογραφικής τους κατάστασης, αλλά όχι μόνο. Ωστόσο, Ανητήρηση υποχρεώσεων από τα κράτη-μέλη ενδυναμώνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα μέτρα αλληλεγγύης. Αντίστροφα, η έλλειψη αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής ευθυνών πλήττει εξίσου την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Με άλλα λόγια, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο αλληλεγγύης εντός του οποίου θα στηρίζονται τα κράτη-μέλη για να βελτιώσουν τα συστήματα ασύλου τους προκειμένου να διασφαλίζεται πλήρως ο σεβασμό των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλων, άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίες, θα εξασφαλίσει ταυτόχρονα την ορθή εφαρμογή του κεκτημένου για το άσυλο και κατά συνέπεια και την ίδια τη λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου. Η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή όπου οι μεταναστευτικές ροές είναι κατά κανόνα μικτές και συμπεριλαμβάνουν μετανάστες, ετούντες άσυλο, πρόσφυγες και ευάλωτα πρόσωπα όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Το λέω αυτό γιατί είναι κρίσιμο να έχουμε πάντα υπόψη μας τον παράγοντα αυτό πως το άσυλο και η μετανάστευση είναι ουσιαστικά διαφορετικές έννοιες με διακριτές ιδιαιτερότητες οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αγνοούνται ή να συχαίονται. Νομίζω πως μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως ο πρωτοφανής αριθμός των ανθρώπων που πνίγηκαν στη Μεσόγειο το 2011 σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να, για να βρουν προστασία είναι μια τραγωδία που δεν θα πρέπει ποτέ να επαναληφθεί. Φυσικά το τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα του ασύλου περιορίζεται από τον κανονισμό του Δουβλίνου που καθορίζει το υπεύθυνο κράτος για την εξέταση αιτήσεων παροχής ασύλου και σχετικά θα ήθελα να τονίσω πως το εν λόγω σύστημα κατανομής θέτει σε μόνιμη βάση τις ανάλογες απαιτήσει σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και δει εκείνα που αποτελούν σημεία εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που αποδυναμώνει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου στο σύνολο του. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις όπου ένα κράτος μέλος δεν δύναται να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις αιτήσει ασύλου που του υποβάλλονται, θα μπορούσαν κατά τη γνώμη μας να εφαρμοστούν οι αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής ευθυνών ως εξής. Τα κράτη-μέλη, οι τοπικές αρχές και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να είναι ενημερωμένοι σωστά σχετικά με τα διάφορα διαθέσιμα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε θέματα ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που σχετίζονται με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Τα συστήματα ασύλου των κρατών μελών πρέπει να αξιολογούνται ανατακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εντοπίζονται καλές πρακτικές ή τυχόν ελλείψεις και να καθίσταται δυνατή και η μετάδοση καλών πρακτικών, αλλά και η εκπόνηση στοχευμένων λύσεων ανταποκρινόμενων σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Πρέπει να ενεργοποιηθούν τα υπάρχοντα ή και να υπάρξουν νέα μέτρα ακόμη, για να στηριχθούν τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν ανάλογες ευθύνες. Εξετάζουμε, παραδείγματο χάρη, τις δυνατότητες που μπορούν να προσφέρουν η κοινή επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου καθώς και η μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Στήριξης για το Άσυλο, ΕΑΣΟ, μπορεί να αποδειχθεί ζωτική σημασία στον λόγο που θέλουμε να δημιουργήσουμε κυρίως μέσω του εντοπισμού ελλείψεως στα συστήματα ασύλου των κρατών μελών, του συντονισμού και της παρακολούθησης της πρακτικής και άμεσης βοήθειας που πρέπει να παρέχεται στα κράτη-μέλη. Εδώ θέλω να υπογραμμίσω τη χρησιμότητα της ανάπτυξης των ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασύλου, αλλά και τον ακόμη πολύ περιορισμένο αντίκτυπο που έχει το ΕΑΣΟ και που πρέπει οπωσδήποτε να αυξηθεί αισθητά στο προσεχές μέλλον η καλύτερη χρήση της συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων κοντιλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα ακόμη βιωτικό, βασικό στοιχείο για τη μετάφραση της αλληλεγγύης σε συγκεκριμένη δράση. Η εισαγωγή οικονομικών κινήτρων για τη μετεγκατάσταση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική σε αυτό το πλαίσιο. Επιτρέψτε μου να τονίσω ξανά ότι κάθε πρόταση και σύσταση που περιέχεται στην έκθεση αυτή στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός πραγματικού χώρου προστασίας, όπου τα δικαιώματα, τα δικαιώματα των ετούντων άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας τηρούνται και προωθούνται δεόντως. Γι' αυτό μερικές προτάσεις είναι οριζόντιες και αγγίζουν επίσης άλλους τομείς της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα συνοριακά μέτρα ή τις πολιτικές θεώρησεις καθώς είναι σημαντικό κάθε πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχεται σε επαφή με την πολιτική ασύλου άμεσα ή έμμεσα να εφαρμόζεται με τρόπο που να σέβεται και να λαμβάνει υπόψη τις υποχρεώσεις μας στον τομέα της διεθνούς προστασίας. Και τέλος αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση τεχνικής φύσεως λόγω υλικοτεχνικών περιορισμών το σχέδιο έκθεσης στην παρούσα μορφή του περιέχει μεν την ουσία όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία τα οποία θεωρούμε ουσιώδη και τα οποία θα προσθεθούν στις τροπολογίες. Φυσικά ενθαρρύνω όλους τους συναδέλφους και δι' τους σκιώδεις εισηγητές να συμβάλλουν στη διαδικασία αυτή και να συζητήσουμε οποιοδήποτε ζήτημα κρίνεται σκόπιμο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλω να συγχαρώ πολύ θερμά τον, τριο... κύριο Τριανταφυλλίδη για τη θαυμάσια έκθεση και για την παρουσίασή του. Περιμένω από μονεσία να κάνω κάποιες συστάσεις μέσω τροπολογιών τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να θέσω μόνο δύο σημεία. Υπό το τμήμα, υπό την ενότητα για την κατανομή των ε, ευθυνών. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης μιλάει για κάποια βασικά σημεία που προτάσει. Ένα από αυτά είναι να βασιστούμε στην εμπειρία, ε, στην εμπειρία του σχεδίου Αρίμα για την εσωτερική επανεγκατάσταση των ετούντων άσυλο που είχε δημιουργηθεί ειδικά για την χώρα μου, για τη Μάλτα. Και όταν ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2011, αυτό το πρόγραμμα είχε επανεγκαταστήσει 227 ετούντες ε, άσυλο από τη Μάλτα σε άλλα 6 κράτη-μέλη. 6 από τα 27. Οκ, καλό. Είναι αλληλεγγύη αυτό. 227 άνθρωποι επανεγκαταστήθηκαν μέσα σε δύο χρόνια νομίζω, σαν να διάστημα δύο ετών, την περασμένη εβδομάδα 275 άνθρωποι φτάσαν στη Μάλτα. Και καμία φωνή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακούστηκε, τίποτα δεν μας, καμία λύση δεν μας βρήκε αυτό το project Γιουρίμα. Οκ, okay, καλό είναι αυτό το project, καλό είναι αυτό το πρόγραμμα, αλλά να μην θεωρήσουμε ότι είναι τόσο επιτυχημένη ιστορία. Νομίζω ότι το project αυτό χρειάζεται πολύ περισσότερα, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα για να θεωρηθεί επιτυχές. Νομίζω ότι όχι μόνο θα πρέπει να επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα, το κάνουμε μόνιμο και να το ανοίξουμε για όλες τις χώρες, όχι μόνο για μία, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει πάνω απ' όλα. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα αυτό δεν λειτουργεί πραγματικά. Δεύτερον, ο εισηγητής λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την οδηγία για την προσωρινή προστασία όταν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πληρούνται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λέει μάλιστα. Όμως, στην κορυφή της κρίσης της Λιβύης, χιλιάδες άτομα άρχισαν να φεύγουν από τη Λιβύη και να φτάνουν στη Λαμπετούζα, Φερρυπίν και στη Μάλτα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τη ζητήθηκε να χρησιμοποιήσει αυτό το μηχανισμό προσωρινής προστασίας μέσω αυτής της οδηγίας. Εκείνη τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε χρησιμοποιήσει διάφορες δικαιολογίες για να μην χρησιμοποιήσει το μηχανισμό. Είπε ας πούμε, α δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί το Συμβούλιο θα το δεχτεί. Από πότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει πρωτοβουλίες με βάση το ότι θα δεχτεί όχι το Συμβούλιο. Ή είπε ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, α δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν υπάρχει μαζική εισρωή χωρίς να προσπαθήσει να προσδιορίσει την αυτή μαζική εισρωή. Ακόμα και για την οδηγία προσωρινής προστασίας θα πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν χρειαστεί, όχι απλώς να τη χρησιμοποιήσει, αλλά να μας πει και πότε και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή, αυτό το κείμενο. Οι σκιώδεις εισηγητές είναι έτοιμοι να εμπλουτίσουν τη συζήτηση. Κυρία Γκυγιόμ, θα προσπαθήσουμε να την εμπλουτίσουμε, Πρόεδρε. Ε, ούτως ή άλλως η έκθεση είναι ήδη ενδιαφέρουσα. Θέλω να χαιρετήσω τον ε, συντάκτη, γιατί ε, αντιμετωπίζει το θέμα του ασύλου και της αγγλικής με τρόπο πολύ πληρή, προτείνει διάφορα μέτρα συγκεκριμένα για να καταλήξουμε σε μια ε, αλληλέγγυα ευρωπαϊκή πολιτική. Τονίζει επίσης το σεβασμό του κοινοτικού κεκτημένου. Μόνο και μόνο γι' αυτό θα άξιζε να το συγχαρούμε. Ε, μπορούμε βέβαια να το συμπληρώσουμε και ξανά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε ως κοιότης εισηγητές. Τρία στοιχεία θα πω για, και μόνο για να σεβαστώ και το χρόνο που μου δίνεται. Πρώτον, για την ε, συνεργασία στην πράξη και κυρίως στο γραφείο, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Σύλλου. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Είμαι σίγουρη ότι το γραφείο αυτό θα πρέπει να έχει τις σωστές ε, να κάνει τη σωστή αποστολή, να αντιμετωπίσει τις ε, προκλήσεις, αλλά για να αντιμετωπίσει και να προωθήσει την ε, αλληλεγγύη θα πρέπει να διερωτηθούμε για τα μέσα που έχει. Μήπως θα πρέπει να του δώσουμε περισσότερα μέσα αυτού του γραφείου. Μήπως να το σκεφτούμε. Επίσης, μέσω τροπολογιών θέλουμε να πούμε ότι η έκθεση θα λέει ότι αυτή η πρακτική συνεργασία να μην υποκαθιστά την ε, νομοθετική εναρμόνιση. Έτσι, υπάρχουν ανεπάρκειες και λήψεις στην νομοθετική εναρμόνιση. Και η συνεργασία στην πράξη δεν είναι αυτή που μπορεί να την αντικαταστήσει την εναρμόνιση. Η αλληλεγγύη είναι επίσης ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ασύλου κοινό, αποτελεσματικό, που προστατεύει τον κόσμο. Και προς το παρόν Έχουμε την αίσθηση σε διάφορες συζητήσεις για το άσυλο και τα κείμενα για το άσυλο ότι οι αναθεωρήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή υποβαθμίζουν τα πράγματα. Για αυτή την νομοθετική λοιπόν εναρμόντιση και για την ε, συνεργασία στην πράξη πρέπει να επαγρυπνήσουμε ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε πιο ενισχυμένη εναρμόνιση. Τελευταίο σημείο για τη συνεργασία και για το θέμα του γραφείου αυτού για το άσυλο θα πρέπει το γραφείο αυτό να συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών εκ του σύνοικης, γιατί είναι θέμα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας και εξαρτάται από αυτή τη συνεργασία. Για την οικονομική αλληλεγγύη, πολύ γρήγορα. Γιατί ούτω ή άλλω έχουμε και άλλε συζητήσει για το Ταμείο, για το Άσυλο και τη Μετανάστευση. Εγώ ασχολούμαι με αυτό. Θέλω να πω εδώ και θα το πω και μέσω μιας τροπολογίας ότι θα πρέπει αυτό το ταμείο να μην είναι υποκατάστατο των εθνικών προϋπολογισμών και η ύπαρξη του ταμείου δεν αποδεσμεύει τα κράτη-μέλη από τις ευθύνες τους και δεν τα απαλλάσσει. Γι' αυτό το σύστημα χρηματοδότησης θα πρέπει να εξασφαλίζει με διαφάνεια ε, την απαραίτητη προστασία. Για το θέμα των ευθυνών και την κατανομή των ευθυνών δεν θα σταθώ. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Αν ε, μπω σε αυτό θα μακρηγορήσω. Για την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Θα κλείσω με αυτή την παρατήρηση. Ίσως είναι το πιο δύσκολο θέμα. Είναι το πιο δύσκολο να το... για να γράψει κανείς γι' αυτό. Η έκθεση του κυρίου Τριανταφυλλίδη είναι πολύ σημαντική όμως, γιατί πραγματικά αντιμετωπίζει αντικειμενικά το πρόβλημα της αμοιβαία δυσπιστίας. Μάλλον περί αυτού πρόκειται και όχι περί αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δουλεύουμε ούτω ώστε να εκφραστεί αυτή η αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη μέσω ενό κοινού, πραγματικά κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου άξιου του ονόματός του. Ευχαριστώ πολύ, κ. Ρωμέβα. Ευχαριστώ πολύ. Διάβαζα με μεγάλη προσοχή την έκθεση. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα για μένα τόσο το σώμα της έκθεσης όσο και η αιτιολογική έκθεση. Είναι πάρα πολύ καλά γραμμένα και τα δύο κομμάτια αυτά και εμείς σαν ομάδα δεν νομίζω θα υποβάλουμε τροπολογίες. Ίσως ε, αν υποβάλαμε κάποιες τροπολογίες θα ήταν απλά και μόνο για να ενισχύσουμε τις ιδέες του εισηγητού. Θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποια στοιχεία σε ό,τι αφορά τα πρόγραμματα επανεγκατάστασης. Αλλά προς το παρόν αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συμμερίζομαι απόλυτα τις προτάσεις. Για δύο λόγους κυρίως. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι προφανές και είναι ένα μήνυμα νομίζω που θα πρέπει και να το μεταφέρουμε ε, σε όσους έρχονται στην Ευρωπαϊκή, ότι ο λόγος που ο κόσμος έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι που μπορούμε να τον Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έρχονται, όχι σε κάποια συγκεκριμένη χώρα. Άρα και η προσέγγιση πρέπει να είναι ευρωπαϊκή. Και θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία όταν αυτό είναι απαραίτητο. Και θα πρέπει να συνεργαστούμε και με τα κράτη τα οποία δέχονται το μεγαλύτερο πληθυσμό. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη και για αλληλεγγύη και για συνυπευθυνότητα. Νομίζω ότι αυτό ακριβώς θέλει να επισημάνει και η έκθεση. Σίγουρα θα μελετήσω ενδελιχέστερα την έκθεση, αλλά προς το παρόν αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συμφωνούμε απόλυτα. Και νομίζω ότι με τις τροπολογίες μας δεν θέλουμε να τροποποιήσουμε, αλλά να ενισχύσουμε την έκθεση αυτή. Κύριε Χίσου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ συνεπτική εκθέση που περιλαμβάνει πάρα πολλά σημεία και με μεγάλη λεπτομέρεια. Νομίζω ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση και νομίζω ότι αποτελεί και αφορμή να συζητηθεί το θέμα αυτό με συγκεκριμένους όρους και να κάνουμε συγκεκριμένη πρόοδο, γιατί το θέμα αυτό το συζητάμε εδώ και καιρό, μιλάμε για θέματα ευθύνης, αλληλεγγύης, αλλά πράγματι εξετάζοντας τη σημερινή κατάσταση, λίγα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Δεν είναι δυνατόν κάποια κράτη-μέλη ε, να κάνουν πίσω, είτε ηθελημένα είτε ακούσια. Θεωρώ ότι αφενός υπάρχει η δυνατότητα μέσω του Ταμείου Ασύλου και ε, Μετανάστευσης να προχωρήσουμε, γιατί είναι και θέμα χρηματοδότησης αυτό. Αυτό την πτυχή λοιπόν θα πρέπει να την καλύψουμε σε ό,τι αφορά μέτρα τα οποία θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν για την ε, βελτίωση της πολιτικής ε, των κρατών μελών, γιατί ξέρουμε ότι κάποια κρατημέλη δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο το οποίο προσδοκούμε, το οποίο επιθυμούμε, ούτε το επίπεδο που απαιτείται από τις οδηγίες. Αφετέρου όμως χρειαζόμαστε και ένα βήμα πέρα από το επίπεδο αυτό. Και δεν είναι νομίζω μυστικό το γεγονός ότι εγώ θέλω να υπάρχει κλίδα πρόσπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. σε ό,τι αφορά την επεξεργασία αιτήσεων ασύλου. Να γίνεται η εξέταση αυτή υπό τακτικούς όρους. Αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για να αφήνουμε μεγάλο ε, ποσοστό των ατόμων αυτών για κάποια λίγα κράτη-μέλη. Θέλουμε ένα κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμαστε Θεωρούμε ότι είμαστε ένας νέος χώρος ελευθερίας, άρα θα πρέπει και στο θέμα αυτό της αλληλεγγύης ε, να το κοιτάξουμε. Πολύ σημαντικό είναι το ότι συμπεριλαμβάνεται και το άρθρο 80 και σε σχέση με τον διάλογο με το Συμβούλιο, το οποίο ως τώρα έχει επιδείξει πολύ διστακτική στάση οι δυσκολίες οι οποίες προέκυψαν στο Δουβλίνο 2 και τις οποίες τις γνωρίζουμε, θεωρώ ότι αποτυπώνονται με πολύ σωστό τρόπο. Θα κάνουμε και μία τροπολογία για να υπάρχει και μία κλίτα κατανομής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να εισαχθεί αυτό άμεσα, αλλά νομίζω ότι αυτό συνάδει και με τις καλές εμπειρίες που μας ανέφερε η Μάλτα. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό. Έχουμε ε, δει ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκύρκοπ. Καταρχάς, Πρόεδρε, Μιλώ όχι από πλευράς ε, Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά από πλευράς της ομάδας σε ό,τι αφορά την, πολιτική, την κοινή πολιτική ασύλου. Έχω μια ελευθερία που δεν θα είχα αν μιλούσα μόνο από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον εισήγητη για αυτό που προσπαθεί να πετύχει. Αλλά σκέφτομαι και το πόσο ελλειπή ήταν η επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ως τώρα σε διάφορους ε, μηχανισμούς, όπως και το Δουβλίνο 1 και 2, σε ό,τι αφορά την απόπειρα κατανομής, αν θέλετε, της ευθύνης για τους ετούντες άσυλο. Τη μοναδική φορά που, τα πετύχαμε, που το πετύχαμε ήταν όταν συμμετείχαμε σε project της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήμουν υπεύθυνο ε, από πλευράς του Ηνωμένου Βασιλείου για την αποστολή στην ε, ε, Βοσνία και ήταν πολύ επιτυχές το πρόγραμμα αυτό σε μια περίοδο κατεπίγουσας ανάγκη στα Βαλκάνια. Και να σας πω ότι δεδομένη και της έλλειψης βοήθειας που έχουμε δώσει στη Μάλτα, στην Ιταλία, σε πρακτικούς όρους, αυτό το μοιραζόμαστε την ευθύνη φαίνεται σχεδόν ειρωνικό Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι ό,τι καλύτερο στον εισηγητή. Ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να προχωρήσουμε με τρόπο που αποτυπώνει, θα αποτυπώνει δίκαια την κατάσταση και τις πιέσεις που δέχονται κάποιες χώρες λόγω γεωγραφικής θέσης. Και ελπίζω και οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Eurodac, τις οποίες θα εξετάσουμε ασφαλώς, θα προχωρήσουν προκειμένου να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε με πιο δίκαιο τρόπο να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα. Κατά τα άλλα, πρέπει να πω ότι καλωσορίζω την πρωτοβουλία από πλευρά τη ομάδα και ελπίζω να είμαστε λίγο λιγότερο εγωιστές σε ό,τι αφορά μεμονωμένες περιστάσεις από ό,τι έχουμε αποδεχθεί στο πρόσφατο παρελθόν. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα έχουν ζητήσει ακόμα κάποιοι συναδελφοί το λόγο. Δύο λεπτά σας παρακαλώ, σας υπενθυμίζω για να έχουμε περιθώρια για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει με τον κύριο Ζιλ Τεκερκόφ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου έχει καταρχάς πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεφλίβη, τον εισηγητή μας για την έκθεσή του. Όντω, είναι πολύ σημαντική η έκθεση. Συμφωνώ με τη δομή και την προσέγγιση που ακολουθεί ο εισηγητής. Αυτή η έκταση μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για όλους μας για το μέλλον, προκειμένου να προσπαθήσουμε σε μια σύντομη χρονική περίοδο, το 2012, να αναπτύξουμε ένα σύστημα ασύλου, το οποίο θα προστατεύει αποτελεσματικά όλους όσοι εκείνοι δικαιούνται άσυλο. Συμφωνώ, όπως είπε ο συγητής, ότι σημαντικό είναι να συζητηθεί η απαραίτητη αλληλεγγύη, η καλύτερη κατανομή, η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να μείνουν μόνο σε θεωρία. Σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποια φάση θα πρέπει όλα αυτά να καταστούν πολιτική, ουσία. Και ως τώρα τα αποτελέσματα δεν ικανοποιούν ασφαλώς στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Πάνω από 120.000 άτομα έρχονται από τρίτες χώρες. Και πολλοί εξ αυτών ετούνται άσυλο παρά το γεγονός ότι δεν το δικαιούνται. Και αυτό συμβαίνει γιατί κάποια κυκλώματα, κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι καταχράζοντας ε, καταχαζόμενοι το σύστημα για, την, ε, το άσυλο, αυτοί θα μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα, χωρίς να εξαναγκαστούν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Άρα, αναφέρομαι σε αυτές τις περιστάσεις, σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει η διαδικασία χορήγησης ασύλου να συνδέεται με ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την ευθύνη την οποία όλοι έχουμε για την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Ό,τι και να κάνουμε στην Ελλάδα. Αν δεν καταφέρουμε να περιορίσουμε την εισρωή μέσω του Εύρου, μέσω της Βόρειας Ελλάδας, μέσω Τουρκίας, ό,τι λοιπόν και να κάνουμε, Αν το πρόβλημα αυτό δεν λυθεί, όλες οι πολιτικές μας και σε ό,τι αφορά το άσυλο θα είναι άκαρπες. Άρα, αυτό ήταν το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω. Και το δεύτερο, και ολοκληρώνω πρόεδρε, είναι το εξή. Όταν παρουσιάζεται μια τέτοια κατάσταση, καταλαβαίνετε συνάδελφοι ότι οι πολίτες της χώρας που έρχεται αντιμέτωποι με το πρόβλημα δεν ε, ικανοποιούνται και αυτοί. Απειλείται ο κοινωνικός ιστός και τελικά αντί να εστιάζουμε την προσοχή μας σε αυτούς που δικαιούνται άσυλο, απειλείται σε πολλές περιπτώσεις η ζωή όλων αυτών των ατόμων. Αυτό φάνηκε και από τις εκλογές στη Γαλλία, από τις εκλογές στην Ελλάδα. Σε κάποιες περιπτώσεις ο κόσμος ε, συμφωνεί και προσεγγίζει ε, ακραίες στάσεις. Και καταλαβαίνετε ότι ασφαλώς εγώ δεν συμφωνώ με μια τέτοια προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρομέρο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η έκθεση του συναδέλφου Τριανταφυλλίδη. Διότι πραγματικά ανοίγει ε, την πόρτα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτή τη διάσταση. Σίγουρα οι χώρε ε, που δέχονται αυτέ τι μεταναστευτικέ πιέσει, τι πιέσει από αυτού του ανθρώπου, ε, χρειάζονται βοήθεια, χρειάζονται υποστήριξη υπάρχουν ε, εμπειρογνώμες. Πολλές φορές ε, μιλάμε και για κάποιες ε, καταχρήσεις, αλλά υπάρχουν εμπειρογνώμονες οι οποίοι εργάζονται σε πολλά μέρη, άρα έχουμε τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για συνεργασία σε αυτό το τόσο λεπτό θέμα. Αλλά, όπως λέει και ο κύριος Τριανταφυλλίδης, το κέντρο, το επίκεντρο είναι ο κανονισμός του Δουβλίνου. Και όσο εξακολουθεί να είναι τόσο ε, επιφυλακτικό το Συμβούλιο, τι να κάνουμε εμείς. Ε, οι χώρες ε, της νότιας όχθης έχουν το πρόβλημα. Οι χώρες της βόρειας όχθης δεν έχουν επίγνωση ότι αυτοί που ζητούν άσυλο δεν το ζητούν για να μείνουν στις χώρες του Νότου, αλλά αυτό που θέλουν είναι να πάνε σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στην Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, αυτοί, αυτές οι χώρες είναι ουσιαστικά οι χώρες ε, προορισμοί και όχι νότια όχθη. Πρέπει λοιπόν ε, να θέσουμε σωστά το, το ζήτημα και νομίζω ότι μόνο αν θέσουμε το πρόβλημα του κανονισμού Δουβλίνου θα τεθεί σωστά το όλο ζήτημα. Πριν από λίγο δυστυχώς μιλήσαμε για αυτή την ε, τραγωδία με αυτό το ναυάγιο αυτού του σκάφους στη Μεσόγειο. δεν έχουμε μόνο αυτά τα τραγικά φαινόμενα. Έχουμε ότι αυξάνεται ακόμη περισσότερο μετά η ζήτηση ασύλου. Και έρχονται κύματα ε, ουσιαστικά όχι από τη Μεσόγειο, αλλά με το αεροπλάνο έρχονται ή ε, δια της Χερσαίας Οδού. Εκεί έρχονται τα περισσότερα κύματα και δεν έχουμε καν στοιχεία το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας και το Τμήμα Μετανάστευσης πρέπει να μας δώσει αυτά τα στοιχεία. Ουσιαστικά η μετανάστευση στην Ευρώπη δεν προέρχεται από τις χώρες Αραβικής Άνοιξης και μιλάμε για τις 10 πρώτες χώρες. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Δεν είναι καμία από αυτές χώρες, χώρα της Νότιας Όχθης της Μεσογείου. Και βέβαια το πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα αριθμών. Μπορεί να μας φαίνεται ε, βέβαια ότι η 200 είναι ένα δράμα και το γιουρίμα ουσιαστικά είναι, τι να πω, γελίων διαστάσεων αν θέλετε. Το πρόβλημα είναι η τραγωδία. Αυτό είναι το ζήτημα, όχι αριθμοί. Οι τραγωδίες που βλέπουμε να συμβαίνουν καθημερινά. Και θα πρέπει να υπάρχουν ε, οι απαραίτητες υποδομές. Θα πρέπει να δούμε πόσα κέντρα κράτησης, ποιοι και πόσοι είναι του ντεσάσιο, τι ανάγκες υπάρχουν αυτή η κατανομή αρμοδιοτήτων, αυτή η αλληλεγγύη, τι ακριβώς συνεπάγεται, τι εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν αντί του κανονισμού του Δουβλίνου, αφού δεν δέχεται το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή να αλλάξει ο κανονισμός του Δουβλίνου. Αυτά τα στοιχεία χρειαζόμαστε. Θέλουμε να προχωρήσουμε, αλλά για να προχωρήσουμε θέλουμε στοιχεία και δεν τα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Ο διευθυντής του Γραφείου Μετανάστευσης ήρθε εδώ και μας είπε δεν έχω στοιχεία για τα κέντρα κράτηση που τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή και στη Μάλτα πράγματι αυτό που είπατε για τον πληθυσμό είναι σίγουρα μια τραγωδία, αλλά περισσότερο μεγαλύτερο ρόλο είναι στην Ελλάδα. Εκεί φτάνουν περισσότεροι. Πώς θα ε, τακτοποιήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να μιλήσουμε έχοντας υπόψη μας όμως γιατί αριθμούς μιλάμε. Και το Συμβούλιο ακόμη, ε, αν πάρει στοιχεία, ίσως να αλλάξει άποψη για το Δουβλίνο και ίσως ε, υπάρξει κάποια επαναχώρηση με τις προτάσεις που γίνονται στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για το άσυλο. Sorry. Ε. Ευχαριστώ. Η κυρία Βίξτρομ έπρεπε να φύγει. Αλλά αυτό μας ε, υπενθυμίζει τη σημασία του σεβασμού του χρόνου. Έχουμε και άλλο σημείο, επαναλαμβάνω, στη ημερήσια διάταξη και μετά έχουμε τη συνάντηση των συντονιστών. Βλέπω και άλλα χέρια να υψώνονται. Θέλετε να μιλήσετε? Θέλετε να πείτε κάτι? Τώρα μπορείτε να μιλήσετε πριν δώσουμε το λόγο στην Κομισιόν και στο τέλος ξανά το λόγο στον εισηγητή τον κύριο Τενταφυλίδη. Ευχαριστώ πρόεδρε που μου δίνετε και εμένα το λόγο. Νομίζω ότι απαραίτητο είναι να κάνουμε μια παρατήρηση πρωτού πάρει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Αυτό που έζησα εγώ στο τέλος της συζήτησης εξακολουθεί να αποτελεί, μάλλον δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σύγχυση ε, μεταξύ της ε, μετανάστευσης ε, των ανθρώπων που θέλουν να βελτιώσουν το βιωτικό τους επίπεδο και τις συνθήκες εργασίας τους σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε η συνάδελφος προηγουμένως, ότι μιλάμε για μετανάστευση και ότι ο κόσμος αυτός που έρχεται στην Ελλάδα δεν θέλει να μείνει στην Ελλάδα, θέλει να συνεχίσει για κάπου αλλού, για τη Γερμανία για παράδειγμα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει τίποτε με τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, με το άσυλο. Εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι όταν πρόκειται για άσυλο, η πρώτη χώρα που μπορεί να χορηγήσει τη βοήθεια, αυτή θα πρέπει να διεκπαιρεώσει την ε, ε, υπόθεση και νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει πολύ γρήγορη διεκπαιρέωση. Αυτοί που λαμβάνουν ε, το καθεστώς ασύλου να βοηθούνται και οι υπόλοιποι που ζητούν, που λένε ότι δεν θέλουν άσυλο, θέλουν να συνεχίσουν για κάπου αλλού, σε αυτούς θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Δεν είναι. Αν θέλουν, μπορούν να επιλέξουν την χώρα που της επιθυμίας τους. Εδώ μιλάμε για γρήγορες διαδικασίες χορήγησης ασύλου και επιστροφής. Εμείς ουσιαστικά νομίζω ότι πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουν ότι στην Ασία για παράδειγμα ε, υπάρχουν οργανώσεις, κυκλώματα τα οποία διοργανώνονται σαν ε, τουριστικά γραφεία. Αυτά δεν έχουν να κάνουν με το άσυλο. Και εδώ θα πρέπει να βάλουμε μια διαχωριστική γραμμή και στη συζήτηση, γιατί ιδάλλως δεν θα προχωρήσουμε. Θεωρώ ότι το Δουβλίνο είναι η σωστή λύση αν υπάρχει σαφής ε, διάκριση μεταξύ μετανάστευσης και ασύλου. Ευχαριστούμε. Κύριε Μπρόνς, γρήγορα πείτε τα είναι μια από τις συζητήσεις όπου τα συμπεράσματα έχουν ήδη προαποφασιστεί. Η δημιουργία ενό κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματο Ασύλου αποφασίστηκε το 2012 ήδη και έχουν αποφασιστεί και τρει πυλώνε του. Άρα δεν έχουμε και πολλά περιθώρια ελιγμό. Δεν ξέρω μήπω θα μπορούσα εγώ με κάποιε υποθέσει κάπω να τάραξω αυτά ε, τα νερά. Αυτοί που ζητούν άσυλο αποφασίζουν για δική του ασφάλεια να φύγουν από τη χώρα διαμονή ή καταγωγή του και να πάνε σε μια χώρα που θα είναι ασφαλή τα εξωτερικά χερσαία σύνορα της Ένωσης ε, δεν θεωρούνται ότι είναι και ε, σε χώρες επικίνδυνες ουσιαστικά. Ούτε είναι και ο τελικό προορισμό των περισσότερων ε, των άσυλο που φτάνουν στην Ευρώπη. Περισσότεροι που ζητούν άσυλο επίσης έχουν παρακάμψει, έχουν διαπεράσει ασφαλέστερες χώρες πριν φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί, ακόμη και αν γνήσια αναζητούν άσυλο, τελικά έχουν μεταμορφωθεί ε, σε οικονομικούς μετανάστες, αν θέλετε, σε μετανάστες επιλογής, αφού έχουν πέρασει την πρώτη ασφαλή χώρα. Αυτοί που δεν είναι γνήσια του ντεσάσυλο πρέπει να ε, επιστραφούν ε, είτε στην πρώτη ασφαλή χώρα που πέρασαν, είτε στην χώρα καταγωγής. του να μιλήσουμε για κοινέ ευθύνε ε, ή καταμερισμό των, επιμερισμό των βαρών αλληλεγγύη είναι περιττό. Δεν υπάρχει βάρος το οποίο χρειάζεται επιμερισμό. Ευχαριστώ πολύ. Επανέρχομαι στον εισηγητή μας τον κύριο Τριανταφυλλίδη. Αλλά νομίζω ότι θέλει το λόγο και Κομισιόν. Γρήγορα, γρήγορα όμως, να μας τα πείτε σύντομα παρακαλούμε. Και μετά θα δώσω στην κύριο Τριανταφυλλη. Θα είμαι σύντομος κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ προς τον εισηγητή για μια ενδελεχέστατη και αρτιότατη έκθεση. Προκατακτικά λίγα είναι τα σχόλιά μου. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Καλωσορίζει το γεγονός ότι το σχέδιο έκθεσης ε, συνολικά στηρίζει την προσέγγιση της Κομισιόν για την αλληλεγγύη και το άσυλο. Δηλαδή, η ευθύνη και η αλληλεγγύη ουσιαστικά είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και θα πρέπει να συμβαδίζουν. Χαιρετίζουμε επίσης την ιδιαίτερα πρακτική προσέγγιση που υιοθετεί ο συγητής σε κάποια πιο συγκεκριμένα ζητήματα που θέτει το σχέδιο έκθεσης. Νομίζουμε ότι πηγαίνουν προς σωστή κατεύθυνση. Τώρα για κάποια τεχνικά ζητήματα μπορούμε να τα συζητήσουμε περαιτέρω και βέβαια με τα χαρά να σας δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια ή υποστήριξη ε, στα τεχνικά ζητήματα για την περαιτέρω ε, βελτίωση της έκθεσης. Υπάρχουν κάποια ζητήματα ουσίας ε, για τα οποία θα ήθελα πολύ σύντομα να κάνω κάποια σχόλια. Η έκθεση για παράδειγμα αναφέρει ότι το Γραφείο Υποστηρίξη θα πρέπει να εντοπίσει ενδεχόμενε αδυναμίε των συστημάτων ασύλου στα κράτη-μέλη θεωρούμε ότι άλλη είναι η δουλειά αυτής της υπηρεσίας της υπηρεσίας ΕΑΣΟ. Βέβαια αυτά θα τα διευκρινίσουμε, μπορούμε να επανέλθουμε. Επίσης ε, είναι προφανέ ότι η έκθεση εκφράζει σαφής ε, ξεκάθαρε επικρίσει κατά του κανονισμού Δουβλίνου. Εγώ δεν μπορώ να ε, παρέμβω αυτή τη στιγμή, καθώ είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσει ε, στην ε, ανακοίνωση για την αλληλεγγύη. Ακολουθήσαμε όμω μια πιο ολιστική προσέγγιση και δεν περιοριστήκαμε στον κανονισμό του Δουβλίνου. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει η αλληλεγγύη να είναι μια ε, συνολική ε, καθολική μέρημνα που θα πρέπει να διέπει όλες τις πτυχές. Σε ό,τι αφορά τώρα τη μελέτη σκοπιμότητας για την κοινή επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και το μόνιμο ε, πρόγραμμα για τη μετεγκατάσταση είναι προτάσει που θα τι εξετάσουμε πολύ προσεκτικά. Τέλο, υπάρχει μια παράγραφο στην έκθεση, στο σχέδιο έκθεση, που λέει ότι οι διαδικασίε επί παραβάση θα πρέπει να θεωρηθούν ω ε, ένα έσχατο μέσο. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, όπω αναμένεται, θα διαδραματίσει πλήρω το ρόλο τη, το ρόλο του θεματοφύλακα των συνθήκων, σύμφωνα με τι υποχρεώσει που τις δίνει η συνθήκη. Πάντω, οι γενικέ γραμμέ μπορούμε να πούμε ότι συμφωνούμε με το σχέδιο έκθεση και πάλι θέλουμε να συγχαρούμε και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τριανταφυλλίδη για την έκθεσή του. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Τριανταφυλλίδη, έχετε το λόγο για να σας ρωτήσετε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο για τον τρόπο που αντιμετώπισαν το το report, το draft report για τα σχόλια που έχουν κάνει. Να τους διαβεβαιώσω ότι οι συνεργάτες μου και εγώ έχουμε σημειώσει όλες τις παρατηρήσεις και ασφαλώς ε, αναμένω τις τροπολογίες οι οποίες θα εμπλουτίσουν ε, την ε, έκθεση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον εκπρόσωπο της Κομισιόν για τα λόγια που έχει πει και οπωσδήποτε είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε στο πεδίο των ε, τεχνικών παρατηρήσεων που έχουν αναφέρει. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Secretariat. Η βοήθεια τους είναι πραγματικά ανεκτήμητη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πληροφορήσω απλώς ότι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι 6 Ιουνίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα είναι στις 10 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μικρόφωνο. Mike, said it right. be out for Πολύ σωστά. Έκλεισε η συζήτηση για αυτό το σημείο. Για τις τροπολογίες η προθεσμία είναι 6 Ιουνίου μέχρι τις 12 η ώρα, όπως είπατε. Θα ανταλλαγούν απόψεις επίσης στις 20 και 21. Για τις τροπολογίες. Η ψηφοφορία στην Επιτροπή μπορεί να γίνει αρχές Ιουλίου. Σας ευχαριστώ όλους. Και τώρα περνάμε στο σημείο για το οποίο ήρθε και ο προσκεκλημένος μας, ο Ζίλντε Κεχκόφα, ο συντονιστής. Τον καλωσορίζουμε θερμά. Καλησπέρα, good afternoon, bon après-midi. Θα γίνει μια συζήτηση για τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση από το συντονιστή για την αντιτρομοκρατία θα παρουσιαστεί από τον Ζήλ Τεκερκόφ. Θα ακούσουμε την παρουσίασή του και μετά θα δώσω το λόγο για ερωτήσεις. Η συζήτηση θα διαρκέσει 45 λεπτά συνολικά. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η συνεδρίαση των συντονιστών. Ο κύριος ε, Ντεκερκόφ έχει το λόγο. Έχετε το λόγο και θα προσπαθήσω να είμαι ε, σύντομος, ώστε να συνεδριάστε και με πολλούς άλλους ε, συντονιστές. Ήρθα εδώ για να μιλήσω για το πρόβλημα των πρόσφατων γεγονότων, αυτό που συνέβη στην Τουλούζη της Γαλλίας, το φαινόμενο του, της όλο τρομοκρατίας. Στη Νορβηγία πριν από ένα χρόνο έγινε ή στη Γερμανία, στη Δανία, ο Ντόλαχαλ στη Σουηδία, στην Ιταλία είχαμε περιστατικά. Όλα αυτά συνοψίζουν δύο εξελίξεις του πάτεν της δημοκρατίας και της απειλής. Καταρχάς, οι μοναχικοί τρομοκράτες, μοναχικοί καβαλάριδες που δεν έχουν να κάνουν μόνο με το τζιχάντ και το δεύτερο, τα ταξίδια που κάνουν Ευρωπαίοι υπήκοοι σε θερμές περιοχές, στο Αφγανιστάν, Πακιστάν πιο παλιά, τώρα όλο και περισσότερο στην Ιεμένη και στη Σομαλία. Δεν είναι σύμπτωση που αυτό το φαινόμενο αυξάνεται. Όπως ξέρετε, ε, η Αλκάιντα δεν μπορεί να κάνει ε, τόσο περίπλοκες επιθέσεις όπως την 19 η Ενάτου, βασίζεται σε υπεργολάβους ε, στην Ιεμένη, στην ε, Σαχέλ και σε, στο Αλσαμπάχ και σε άλλες ομάδες. Ε, και με μεγαλύτερη, όλο και μεγαλύτερη ανησυχία βλέπουμε τις εξελίξεις στην Αφρική. Ο εφιάλτης θα ήταν η QIM και διάφορε ομάδες στη Σαχέλ να συνεργαστούν. Είδατε στο βόρειο Μαλί της εξελίξεις, Μποκουαχάμ στη βόρειο Αλγερία και Σομαλία. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ε, δεν υπάρχει μόνο υπεργολαβία. Η Αλκάιδα προσπαθεί να ενθαρρύνει μέσω μιας προπαγάνδας τοχοθετημένης τους δυτικούς να δράσουν όπου και όταν μπορούν ακόμα και σε μικρή κλίμακα και να υποφεληθούν από κάθε ευκαιρία που έχουν για μικρές επιθέσεις. Αν διαβάσετε τις ε, πρόσφατες δημοσιεύσεις, ακριβώς αυτό το μήνυμα προσπαθεί να περάσει η Αλκάιντα. Φυσικά, αυτό είναι μια τεράστια πρόσκληση για την ε, όσο ασχολούνται με, και βρίσκονται στην υπηρεσία πληροφοριών. Είναι δύσκολο να του εντοπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς τους μοναχικούς ε, καβαλάριδε, την έβριση την αντλούν. Δεν, δεν τους έρχεται έτσι ξαφνικά, αλλά δρούν μόνοι τους. Και γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολη η αντιμετώπιση τους. Είμαι λοιπόν ευγνώμων προς αυτή την Επιτροπή που θέλει να ψάξει αυτό το θέμα για να δει τι μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο φαινόμενα. Τώρα, θα ήθελα να στραφώ σε αυτά τα δύο φαινόμενα, στους μοναχικούς καβαλάδε και στους ταξιδιώτες. Η σημερινή στρατηγική είναι επαρκής για να αντιμετωπίσει την σόλο τρομοκρατία θα έλεγα ναι, ότι η στρατηγική που υιοθετήσαμε το 2005, ναι, είναι ακόμα επίκαιρη. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα σε, διάφορες, σε διάφορα επίπεδα. Καταρχά σε επίπεδο πρόληψη. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να αυξήσουν την συνείδηση και την αφύπνιση όλων εκείνων που μπορούν να εντοπίσουν ε, όσο και πιο νωρί γίνεται σημάδια ρίζος, παστικοποίησης, ε, Μιλάμε για γονείς, για δασκάλου, ακόμα και για ανθρώπους που δουλεύουν ε, στον τομέα της υγείας. Γιατί ε, ξέρετε ότι δύο από αυτού είχαν σοβαρά ε, προβλήματα ψυχικά. Και οποιαδήποτε πληροφορία ή οτιδήποτε έχουν εντοπίσει να το διαμηνήσουν στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, ε, η κατάρτιση τη αστυνομία που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η βελγική αστυνομία έχει μια σημαντική εμπειρία από την αστυνόμευση των κοινοτήτων. Έστειλαν δηλαδή ένα εγχειρίδιο ε, στους αστυνομικούς ε, για το πώς μπορούν να ανοιχνεύσουν πολύ νωρί σημάδια ρίζοσπαστικοποίησης. Πολύ περισσότερα πρέπει να γίνουν σε αυτό το επίπεδο. Ένα άλλο σημαντικό μήνυμα είναι να αυξήσουμε την αντοχή των ευπαθών κοινοτήτων για την επόμενη μέρα. Και αυτό είναι το βασικό μάθημα από τις πρόσφατες επιθέσεις. Γιατί δεν μπορούμε να αποτρέψουμε όλες τις επιθέσεις. Αποκλείεται να εξασφαλίσουμε 100% ε, επίθεση. Να... Θα πρέπει λοιπόν ε, πολύ νωρίς να ενημερώσουμε τις κοινότητες, ούτως ώστε να μειώσουμε την αναπόφευκτη πόλωση που θα προκαλέσει μια τέτοια μεγάλη επίθεση. Ε, με μεγάλη χαρά ήταν στη Γαλλία, ας πούμε, ότι οι επικεφαλής της α, μουσουλμανικής κοινότητας μαζί αντέδρασαν στα γεγονότα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι το ίντερνετ φυσικά. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το ίντερνετ παίζει σημαντικό ρόλο, όχι μόνο εμπνέοντα ε, και βοηθώντας αυτή τη διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης, αλλά και στην ε, εκτέλεση αυτών των επιθέσεων. Πρέπει να έχουν τεράστια πράγματα εκεί. Ξεκινήσαμε, αλλά δεν αρκούν αυτά που κάναμε. Αυτά που κάναμε. Καταρχάς παρακολούθηση του ίντερνετ, επίσης ε, στο σελίδες να φεύγουν, να τις κατεβάζουμε και η χρήση του ίντερνετ με ενεργητικό τρόπο, ούτω ώστε να έχουμε και την άλλη ιστορία, την αντίθετη. Ε, θα ξέρετε ότι η Europol έχει αναπτύξει ένα project, Check the Web λέγεται, όπου η Europol προσπαθεί να, προσπαθεί να συλλέξει τα προϊόντα που προκύπτουν από τη διαδικασία ε, εποπτεία των κρατών μελών. Αυτό είναι το παθητικό επίπεδο. Η Europol δηλαδή συλλέγει αυτά που τον καρπόστον της παρακολούθησης των κρατών μελών. Χρήσιμο θα ήταν η Europol να είναι και πιο δραστήρια, πιο ενεργητική. Να κάνει δηλαδή ίδια κάποια πράγματα. Έχει ούτως ή άλλως ομάδες με καλούς εμπειρογνώμονες για αυτό το θέμα. Ε, όχι μόνο σε παθητικό επίπεδο στο ίντερνετ, αλλά ε, να ελέγχει το ίντερνετ, check the web, να ψάχνει τα blog, τα κοινωνικά δίκτυα με πιο ενεργητικό τρόπο. Έτσι. Δεύτερον, κατεβάζουμε τις παράνομες ιστοσελίδες. Ευαίσθητο θέμα, το ξέρουμε. Η Κομισιόν ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια ένα διάλογο με την ESP, αλλά όχι πολύ θερμό. Ούτως ώστε να υπάρξει μια τέτοια δράση Πρέπει να ενισχύσουμε αυτό το διάλογο. Υπάρχει ένα project ε, με ηγετικό ρόλο της, την Ολλανδία με τίτλο «Καθάρισε το ίντερνετ». Πρέπει να την υποστηρίξουμε. Τρίτον, πιο ευαίσθητο, να χρησιμοποιούμε το ίντερνετ ούτω ώστε να περνάμε και μια άλλη ε, λογική μέσα από αυτό. Ε, την αντίθετη λογική, αν θέλετε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε, αν θέλετε, τις προϋποθέσεις μέσα ε, από τις οποίες όσοι θέλουν να στέλνουν τέτοια μηνύματα, αντίθετα από τα τρομοκρατικά, μπορούν να το κάνουν. Ακόμα και να μεταφράζουμε, αν θέλετε, κάποια πράγματα. Ε, ίσως κάποια πράγματα που υπάρχουν στο ίντερνετ στα αραβικά, αλλά όχι στα αγγλικά, καλό θα ήταν να το κάνουμε. Επίσης, οι φυλακές. Ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί είναι φυτόρια ε, παραγωγής ριζοσπαστών. Αρχίσαμε μια δουλειά, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερο όμως εκεί με πρωτοβουλία της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας. Έχουμε ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που ε, διαχειρίζονται τις φυλακές να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Ε, το πρόβλημα της ε, ριζοσπαστικοποίησης στη φυλακή. Πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα. Οι φυλακές, ε, οι φύλακες και οι υπηρεσίε πληροφοριών πρέπει να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα για την κατάρτιση του, των φυλάκων, Πρέπει να εποπτεύουμε επίσης κάποιους ανθρώπους που αποφυλακίζονται για κάποιο διάστημα. Επίσης η επίθεση της Τουλούζης θέτει ξανά το θέμα της διαθεσιμότητας μικρών όπλων και εκρηκτικών. Ε, το Συμβούλιο, όπως ξέρετε, ολοκληρώνει τις διαδικασίες διαπραγμάτευσης για τον καονισμό, για τις πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών. Είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση. Νομίζω εγώ δεν είχα την εμπειρία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η σημερινή νομοθεσία για τα μικρά όπλα και να δούμε αν πρέπει μήπως να λάβουμε μια νέα απόφαση ή να κάνουμε νέες ε, προτάσεις, ούτως ώστε να γίνει πολύ πιο δύσκολο να βρίσκει κανείς ε, μικρά όπλα. Για τους μοναχικούς καβαλάριδες. Αυτά. Τώρα, για, την, ε, για τα ταξίδια που κάνουν διάφοροι τζιχάντιστς, διάφοροι τρομοκράτες, υπάρχουν πολλές προτάσεις. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο λίγες. Καταρχά, θα ήθελα να προσκαλέσω τη Europol και τη Frontex. Η Frontex, όπω ξέρετε, από την υιοθέτηση του νέου κανονισμού είναι σε θέση να συλλέγει προσωπικά δεδομένα ε, στα πλαίσια των επιχειρήσεών τη. ούτως ώστε να κάνουμε να κάνει μια κοινή έκθεση για τους τρόπους, ε, τα μέσα μεταφορά, το modus operandi, ε, το δίκτυο διευκόλυνσης. Πού πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ε, ποια, ποιες είναι ποια είναι αυτά τα θερμά σημεία. Το PNR είναι μία λύση, δεν είναι η πανάκια, είναι ένας τρόπος για να α, δούμε αυτούς τους, να παρακολουθήσουμε αυτούς τους ύποπτους ταξιδιώτες. Παραδείγματος χάρη ο τύπος που προσπάθησε στην Times Square να, πριν από κάνα δύο χρόνια να προκαλέσει την έκρηξη ενός αυτοκινήτου. Πήγαινε στο, τα προηγούμενα χρόνια στο Πακιστάν. Ε, έκανε τέτοια επίθεση στο Πακιστάν. Θα μπορούσε αυτό να μα σημαίνει ένα καμπανάκι, έτσι, για το πώ ε, λειτουργεί το επίπεδο τη πρόληψη. Μια τρίτη πρόταση, ε, κάτι που έχω πει κατ' επανάληψη και είδα ότι ο πρώην πρόεδρο τη Γαλλία έκανε την ίδια πρόταση. Ε, καλό θα ήταν να τροποποιήσουμε την νομοθεσία για την τρομοκρασία, την απόφαση πλαίσιο που υιοθετήθηκε το 2002 και τροποποιήθηκε το 2008, ούτω ώστε να ποινικοποιήσουμε το ταξίδι στο εξωτερικό για να πάει κανεί σε ένα στρατόπεδο εκπαίδευση έχουμε ε, επεκτείνει τον ορισμό για να καλύψουμε και την ε, κατάρτιση, τη διδασκαλία, ε, την δημόσια πρόκληση. Δεν αρκεί αυτό, αλλά πρέπει να υπάρξει και αστομική συνεργασία με τις αρχές αυτών των χωρών. Επίσης, να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες, με τις χώρες διέλευσης, με τις χώρες προορισμού. Ορισμένες χώρες Προφανώς έχουν πληροφορίες. Θα πρέπει να δώσουμε τεχνική αρρωγή σε αυτές τις χώρες και να τις βοηθήσουμε να ανοιχνεύουν στα σύνορα τους ύποπτους ταξιδιώτες, τους ύποπτους επιβάτες. Εκεί μπορούμε να παίξουμε σημαντικό ρόλο. Αυτά προσπαθούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το Πακιστάν, την Αφρική, τη Σαχέλ με επιπλέον μέσα για να ενισχύσουμε το δυναμικό απόκρισή τους. Αυτά με δύο λόγια. Κάποιες συμβουλές που έδωσα στους Υπουργού στο γεύμα στο πλαίσιο του τελευταίου Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο. Προσπαθήσαμε να δουλέψουμε σε αυτά διάφορα επίπεδα, αλλά απόκειται στην Κομισιόν και στην ε, ΕΑΣ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, να ολοκληρώσουν την προσπάθεια. Σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή κάποιον από των πιο δύσκολων ζητημάτων στη διαχείρισή τους. Να ζητήσω από όλα τα μέλη που ζήτησαν το λόγο να κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι όσο πιο συνοπτικοί γίνονται, γιατί ήσασταν και εσείς το ίδιο συνοπτικό στην παρουσίασή σας, η κυρία Φλότρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλή σας ημέρα ε, κύριε Ντικερκόφ. Το θέμα το οποίο με απασχολεί είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συγκροτήθηκε μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά σκεφτόμαστε και πανεξετάζουμε τις πρακτικές και τις πολιτικές ε, που έχουμε χαράξει για την ε, καταπολέμηση της δημοκρατίας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά και τον τρόπο δράση ε, των υπηρεσιών πληροφοριών και των μυστικών υπηρεσιών και Ιδίω αυτά που έγιναν στη Γαλλία, μας ε, δημιουργούν πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Σίγουρα διαφορετική είναι η προετοιμασία ανάλογα με τη χώρα. Είπατε κι εσείς ότι υπάρχει ρίζος παστικοποίηση με ε, μοναχικών εκτελεστών. Ε, όμως ο συγκεκριμένος κύριος ε, τον παρακολουθούσαν οι μυστικές υπηρεσίες. Πριν από κάποιους μήνες είχε και ένα ραντεβού με τις μυστικές υπηρεσίες ε, κάποιους μήνες πριν από τις φρικτές αυτές επιθέσεις και ο πρώην διευθυντής ε, της υπηρεσίας ασφάλειας, ο κύριος Μπονέλ, εκπλήσεται ε, γιατί ο κύριος αυτός είχε και κάποια αλληλογραφία με τις υπηρεσίες ε, ε, ή κάποιον ανταποκριτή και δεν ξέρουμε ακριβώς. Δηλαδή κάποιος που ίσως τον χρησιμοποιούσαν οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας στον αγώνα καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Και στράφηκε κατά τον αυτών για τους οποίους υποτίθεται ότι εργαζόταν. Ε, επομένως η υπόθεση του Μεράχ στη Γαλλία ε, ανοίγει πάρα πολλά θέματα. Ε, δεν ξέρω κατά πόσον πρέπει να δημιουργήσουμε, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τα μέσα τα οποία υπάρχουν. Επίσης ξέρουμε ότι με ρευστά είχε προμηθευτεί παράνομα όπλα πάνω από 20.000 ευρώ αξίας και μετά την πρώτη ε, από κατά των στρατικών στόχων δεν επιλήφθηκε στρατοδίκης, ε, δεν ε, πήγε πολύ καλά η έρευνα, κάτι που δεν έπρεπε να γίνει δίνονταν στοιχεία κάθε πέντε λεπτά, παντού όλοι τα ήξεραν τι γίνεται και επίσης ουσιαστικά τον ε, έκαναν σουρωτήρι από τις σφαίρες οι άντρες της αντιτρομοκρατικής. Δεν μπορώ να πω ότι ε, είναι ικανοποιητικό ο τρόπος με τον οποίο ενήργησαν τα, όλες αυτές οι υπηρεσίες και οι, οι δυνάμεις ασφαλείας. Ε, ούτε τα μέσα που πήγαν στη διάθεσή τους τα αξιοποίησαν με τον σωστό τρόπο. Επομένως θα πρέπει ο καθένας να θέσει τα ερωτηματικά του και να θέσει και τις απαιτήσει του για το ποιες είναι οι δυνατότητες ελέγχου αυτών των υπηρεσιών πληροφοριών. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να, να δω είναι εσάς αν σας ενδιαφέρει όλη αυτή η υπόθεση του ΜΕΡΑΧ, του, του, του δράστη της Τουλούζης, ε, και τι συμπεράσματα μπορούμε να συνάγουμε. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για την αξιοπιστία, για το κύρος των πολιτικών κατά της τρομοκρατίας. Ε, μπορούν οι πολίτες να εμπιστεύονται τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γιατί από αυτό θα κρυφθεί και επιτυχία ε, όλη αυτή τη προσπάθεια. Εδώ δυστυχώ νομίζω ότι έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα στη διάθεσή μα, τα οποία μα δημιουργούν ερωτηματικά πολύ ξεκάθαρα και θίγουν, πλήττουν αυτήν την εμπιστοσύνη και στις πολιτικές που εσείς ε, συντονίζετε εξ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίρκερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κέρκχοφ για την παρουσίαση των προβλημάτων και των στρατηγικών που μας παρουσιάσατε. Κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη, για τις δραστηριότητες της Αλκάιντα στην ζώνη Σαχέλ που φαίνεται ότι είναι εξαιρετικά επιτυχής και επηρεάζει και τα πολιτικά δρόμενα. Από τις αναλύσεις σας προκύπτει ότι υπάρχουν τεκμήρια ότι τα χρήματα τα οποία αποτελούν έσοδα από το εμπόριο ανθρώπων τα διαχειρίζονται η Αλκάιντα στη Σαχέλ για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Δεν το ξέρω για το κατά πόσον, το κατά πόσον έχουν γίνει σχετικές αναλύσεις. Εγώ έλαβα πληροφορίες βάσει των οποίων φαίνεται ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τα πράγματα, ότι από ό,τι φαίνεται αυτό μάλλον θα μας οδηγούσε να κάνουμε πιο έντονους ελέγχους και για τα κυκλώματα διακίνησης. Δεύτερη ερώτηση για τους μεμονωμένους αυτούς δράστες σύμφωνα με την εμπειρία σας και τις αναλύσεις σας, υπάρχει όλο και μεγαλύτερη τάση να είναι ευρωπαϊκή η προέλευση των μεμονωμένων αυτών δραστών που δεν είχαν στο παρελθόν τίποτα να κάνουν με το Ισλάμ και τον Ισλαμισμό. Και πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να υποπτεύουμε ομάδες που προσελκύουν, προσελτίζουν και εκπαιδεύουν στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν τέτοια άτομα. Τρίτη ερώτηση. Είπατε ότι η Europol θα πρέπει να είναι πιο δραστήρια, proactive. Θα μπορούσαν να γίνουν και έρευνες ε, συγκαλυμμένων με φορέων. Και στο πλαίσιο αυτό μπορείτε να φανταστείτε συνεργασία, πιο στενή συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών προκειμένου να ε, στεφτούν με επιτυχία τέτοιε δράσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σκυρκόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω για έναν άλλο τομέα, αν μου επιτρέπετε, γιατί δεν έχω και πολύ μεγάλη ε, γνώση. Ε, τι Δεν θέλω να ξέρω όλε τι πληροφορίε για το τι κάνουν οι υπηρεσίε πληροφοριών για να προστατεύσουν εμένα, την οικογένειά μου και του πολίτε τη χώρα μου ή τη Ευρώπη. Αλλά θέλω να είμαι ικανοποιημένο για το ότι υπάρχει κάποιο έλεγχο ε, τη δράση του. Και αυτό ο έλεγχο να βασίζεται στο κοινοβουλευτικό σύστημα. Σε διάφορε χώρε οι υπηρεσίε ε, πληροφοριών έχουν ε, να λογοδοτήσουν σε κάποια κοινοβουλευτική επιτροπή. Υπάρχουν λίγοι άνθρωποι που ε, εκ μέρου του Κοινοβουλίου της χώρας αλλά και των πολιτών φροντίζουν οι υπηρεσίες αυτές να λειτουργούν ε, τηρώντας κάποιους κανόνες, λογικούς κανόνες. οι τρομοκράτες ε, δεν μας ε, διαφημίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα δράσουν. Ε, είναι διαφορετικοί ως προσωπικότητες και έχουν και διαφορετικούς τρόπους δράσης, αλλά αυτό που τους ενώνει κατά κάποιο τρόπο είναι ότι δεν έχουν καμία, κανένα δισταγμό να σκοτώσουν, να αφαιρέσουν μια ανθρώπινη ζωή. Εμείς θέλουμε να ζήσουμε όμως ειρηνικά και θέλουμε και οι αρχές επιβολής του νόμου να μας εξασφαλίζουν την προστασία. Το ίδιο θέλουμε και από τις υπηρεσίες ε, πληροφοριών. Έχετε να σχολιάσετε κάτι πάνω στο τι παραπάνω θα μπορούσε να γίνει, ώστε να υπάρχει αυτός ο βασικός έλεγχος. Αυτό είναι το επιδιωκούμενο, αυτό είναι το ζητούμενο. Υπάρχει αυτός ο βασικός έλεγχος σε κάθε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι υποχρεώσεις υπάρχουν, αν δεν υπάρχει αυτός ο έλεγχος, για να τον θεσπίσουν οι χώρες. Ευχαριστώ κύριε Λάτφορτ. Θα ήθελα ακριβώς πάνω σε αυτό και εγώ να εκφέρω τις απόψεις μου, γιατί και εμένα με ενδιαφέρει το ζήτημα ιδιαιτέρως Η λυπηρή συνήθεια των υπηρεσιών πληροφοριών και των κυβερνήσεων να επικαλούνται ε, κατά ρουτίνα το απόρριτο, την ανάγκη για ηχεμή όταν γίνεται μια έρευνα, Εντάξει, φυσικά έχουμε ότι υπάρχουν γνήσια ζητήματα ε, ασφαλείας, τα οποία σχετίζονται με τις μεθόδους, με τους πληροφοριοδότες και σίγουρα όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να παραμένουν απόρριτα, να παραμένουν εμπιστευτικά. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε κάθε συμφέρον και ενδιαφέρον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε ένα μοντέλο κοινοβουλευτικού ελέγχου αυτών των υπηρεσιών πληροφοριών. Αυτό θα μας δώσει ακριβώς ε, την ε, εμπιστοσύνη σε αυτές τις υπηρεσίες, ότι όχι μόνο μας προστατεύουν, αλλά τηρούν και τις δεσμεύσεις για την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο στο Ηνωμένο Βασίλειο που την κυβέρνηση σας αυτήν την εβδομάδα κατατέθηκε την Επιτροπή ε, Ασφαλείας θα την κάνει πραγματικά κοινοβουλευτική και δεν θα αναφέρεται στον Πρωθυπουργό, αλλά στο Κοινοβούλιο. Χαίρομαι που η συντηρητική κυβέρνηση έκανε κάτι που δεν έκανε ποτέ η κυβέρνηση των εργατικών, τέλος πάντων. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα. Κύριε Τεκεκόφ γνωρίζετε και η Ελέν Φλότρ και εγώ προσωπικά και άλλοι έχουμε ξαναφέρει στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα της πλήρους λογοδοσίας και ευθύνης ε, των ε, υπηρεσιών πληροφοριών που καλύπτονται κατά κάποιο τρόπο από τις κυβερνήσεις και πολλές φορές ε, έχουν συνενοχή σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και βασανισμού ανθρώπων. Εγώ δεν θα σταματήσω ποτέ να μάχομαι για να υπάρχει πλήρης λογοδοσία αυτών των υπηρεσιών. Μιλήσατε επίσης για τη χρήση των στοιχείων ε, των δεδομένων επιβατών, PNR, για ένα πιο αποτελεσματικό profiling. Πριν από τρία χρόνια ήμουν εισηγήτρια στο κοινοβούλιο εδώ για μια έκθεση και είχα πει ότι ή πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι και να πούμε ότι ουσιαστικά πρόκειται για profiling, να το πούμε ξεκάθαρα, και όχι ότι απλά κάνουμε έτσι μια μελέτη συμπεριφοριστική, συμπεριφοριστικού τύπου, για να εντοπίσουμε πιθανούς κινδύνους. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν να έχουμε κάποια αντίδραση. Είπατε εσείς. Υπάρχει κάποιος που πάει στο Πακιστάν ε, κάθε χρόνο για δύο εβδομάδε και ξαφνικά πάει και μένει έξι μήνες. Αυτό μπορεί να είναι ύποπτο, μπορεί και να μην είναι. Μπορεί να έχει την άρρωστη μητέρα του εκεί και γι' αυτό να πήγε και να μείνει έξι μήνες και να από τη εκλογική περιφέρεια. Δεν είναι αθέμητο να τον ε, ελέγξουμε, αλλά αθέμητο είναι να κρατήσουμε τα στοιχεία για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί αυτό σημαίνει φακέλωμα. Και εγώ νομίζω ότι πρέπει να σβήνουμε οποιοδήποτε ίχνος αυτή τη σημαία ε, ε, ότι δείξαμε ενδιαφέρον για συγκεκριμένο άνθρωπο, εφόσον βέβαια αποδέχθηκε ότι δεν συνέτρεχε λόγο. Ο κίνδυνο αυτού του profiling του φακελώματο κατά κάποιο τρόπο δεν είναι μόνο ότι κάποια μηχανήματα θα παίρνουν σε αυτόματε αποφάσει για το ποιο είναι υποπτό ή όχι. Αλλά ίσω κάποιο έχει κάποιε συνήθειε όταν ταξιδεύει και γι' αυτό ε, κριθεί ότι πρέπει να ε, τον διπλοτσεκάρουμε, ενώ δεν υπάρχει τίποτα ύποπτο σε αυτόν. Και αυτά τα άτομα θα στιγματιστούν και θα τους ακολουθεί αυτή η ρετσινιά χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Πώς θα μπορούσαμε αυτό να το αποφύγουμε. Ευχαριστώ. Κυρία Χιμένες Σερίλ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Μιλήσατε για το μοναχικό τρομοκράτη και για τον ε, τζιχαντιστή τρομοκράτη. Ήταν πολύ σαφής ε, η παρουσίασή σας και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας όταν μιλάτε για πρόληψη και για την ανάγκη να ανοιχνεύσουμε, να εντοπίσουμε την ριζοσπαστικοποίηση με ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης πληροφορίες ε, μέσω της αστυνομίας. Πράγματι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε εντελώ τι τρομοκρατικέ επιθέσει, μπορούμε όμω πολλέ από αυτέ να σταματήσουμε. Και γι' αυτό χρειάζεται καλύτερη επικοινωνία. Πολλέ φορέ ε, πολλοί κόσμοι δεν γνωρίζει τι γίνεται για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και έχει κάποιε προκαταλήψει και γι' αυτό είναι πάντοτε κατά. Ε, θα ήθελα να μου πείτε επίσης αν η παρακμή ε, της Αλκάιντα για την οποία μιλήσατε θα οδηγήσει και σε μείωση της τρομοκρατίας ή αν έχουμε απλά μία μεταμόρφωση, μία, ένα μετασχηματισμό της τρομοκρατίας. Ε, υπάρχει και ένας άλλος, ε, ε, μια άλλη μορφή τρομοκρατίας, η αυτονομιστική τρομοκρατία, η ΕΤΑ για παράδειγμα είναι μια τέτοια τρομοκρατική οργάνωση. Όταν έχουμε εκθέσει από τη Europol που βεβαιώνουν ότι εξακολουθούν να, να έχουν όπλα αυτοί οι, οι, οι άνθρωποι γιατί είδαμε ότι υπήρξαν και κάποιες κατασχέσεις ε, και κάποιες συλλήψεις ε, και χθε στην ε, Ισπανία και τη Γαλλία Συνελήφθησαν δύο συγκεκριμένα ηγετικά στελέχη της ΕΤΑ, οι οποίοι ήταν ένοπλοι και μάλιστα είχαν και κρυκτικά έτοιμα για να διαπράξουν κάποια επίθεση. Άρα, όταν λέει η ΕΤΑ ότι έχει πλέον καταλήξει και χειρία, μπορούμε να την πιστέψουμε. Τι εξοπιστία έχει η ΕΤΑ. Ευχαριστώ πολύ να επιδράσετε και να συνοψίσετε τις απαντήσεις σας, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρία Φλότρα, για τη Φερμέρα. για την υπόθεση Μεράχ και για τα θέματα που μπαίνουν εκεί. Ε, σωστές ερωτήσεις. Η κατάσταση είναι η εξή. Το κείμενο των συνθήκων όπως έχει σήμερα στον τομέα των πληροφοριών λέει ότι αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ε, το άρθρο 4 το αναφέρει αυτό ρητά. Μπορούμε να πούμε διάφορα πράγματα, αλλά δεν έχουμε αρμοδιότητα για να παρισφρήσουμε εκεί. Είναι επιλογή των κρατών μελών. Μπορούμε να, το, να λυπηθούμε που έγινε αυτή η επιλογή, αλλά έτσι είναι. Τα ερωτήματα που θέτεται είναι σωστά ερωτήματα και θα ήταν ενδιαφέρον όταν γίνουν αυτές οι κυβερνητικές αλλαγές στη Γαλλία, να δούμε τι λειτουργήσε και τι δεν, και τι δεν λειτουργήσε. Πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να βγάλουμε τα διδάγματά μας. Ε, αυτές είναι κάποιες ε, περιπτώσεις που αναφέρονται μεταξύ πολλών. Τώρα, αν αποδειχθεί ότι υπήρξαν ε, ελλείψεις στο μηχανισμό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μηχανισμό, έτσι. Απλώς ε, καθώς αλλάζει η τρομοκρατική συμπεριφορά, εμείς θα πρέπει να κινηθούμε προς κάποιες από τις κατευθύνσεις που ανέφερα και να εξελιχθούμε επίσης για το ερώτημα που θέσατε για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και ο κύριος Κέρκοπ και η Σάρα Λάντφορντ το, έθεσαν το ίδιο ερώτημα. Φυσικά και εγώ είμαι θειασότης ε, εθνικών κοινοβουλευτικών ελέγχων. Και όταν το συζητήσαμε, νομίζω ότι μια ιδέα είχα πει ότι μια ιδέα θα ήταν να δικτυώσουμε τις ε, αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές ε, των κρατών μελών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, για να δούμε τι, ποιες είναι οι καλές πρακτικές. Παραδείγματο χάρη, ξέρω το βελγικό μοντέλο, όπου το κοινοβούλιο ε, βασίζεται σε άτομα που ασχολούνται με τον έλεγχο και ενημερώνουν την καθήλυνα αρμόδια επιτροπή. Για τον έλεγχο των αστυνομικών, μερικές φορές είχαμε σκεφτεί να υπάρξει δικτύωση όλων των αστυνομιών της Ευρώπης, ας πούμε. Ε, και να κάνουμε... Θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, ας πούμε, στην Ευρώπη. Και τα κράτη που δεν έχουν κάτι τέτοιο θα μπορούσαν ε, να, να το κάνουν. Επίσης, προσπάθησα πίσω πείσω τους ε, συναδέλφους της Κομισιόν και της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Πρέπει να βοηθήσουμε και τις χώρες της Νοτιού Μεσογείου, της Αραβικής Άνοιξης, με τις οποίες μπορούμε να επικρίνουμε ως προς το πώς δούλευαν στο παρελθόν τα παλιά ε, καθεστώτα δηλαδή. Ε, αλλά μπορούμε να τις βοηθήσουμε. Προφανώς ε, οι υπηρεσίες αυτές, οι μυστικές και οι υπηρεσίες προφοριών διαλύθηκαν για λόγους κατανοητούς. Αλλά πρέπει να τις βοηθήσουμε τώρα. Εδώ μπαίνει ένας ρόλος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενθαρρύνουμε αυτές τις χώρες να δημιουργήσουν έναν κοινοβουλευτικό έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ε, προφοριών. Τώρα για το ερώτημα για το Μαγκρέμπ, ε, τον Ισλαμισμό στον, στο Μαγκρέμπ και τον τρόπο χρηματοδότησης για τη σωμα, σωματεμπορία, για τα λίτρα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα λίτρα χρηματοδοτούν... Ε, υπάρχουν απίστευτα ποσά. Επίσης όμως και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Και εγώ είδα πολλές εκθέσεις που μιλάνε για διαφορετικά πράγματα, για την ε, ε, τη συμμετοχή της ομάδας ΑΚΜΗ και στην ε, διακίνηση της κοκαίνης, παρότι δεν κάνουν οι ίδιοι κοκαίνη, ας πούμε, διακίνηση κοκαίνης, εποφελούνται και παίρνουν λεφτά. Για την σωματεμπορία, τη σωμα... το εμπόριο ανθρώπων, ήταν μία από την πρώτες που έκανα. Ζητάω από τη Frontex και τη Europol να αναλύσουν αυτό το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπινων όντων. Τώρα, αν οι ομάδε στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν επίτηδε προσπαθούν να προσελκύσουν Ευρωπαίου, η απάντηση είναι προφανώ ναι. Ο Μέρα πήγε όμω από μόνο του. Έκανε μια απίστευτη διαδρομή, μια Οδύσσια. Πέρασε από την Αίγυπτο, από την Ιορδανία κτλ. Και έφτασε στο Πακιστάν. Ήταν ικανός όμως, γιατί δεν πήγε στις ε, ζώνες που ζουν οι διάφορες φυλές. Πήγε στην καρδιά όμως της τρομοκρατίας στο Πακιστάν μερικές μέρες και έμεινε και κοντά στο Ισλαμαμπάντ. Εκεί ε, καταρτίστηκε έτσι στο πώς να χειρίζεται τα όπλα. Ε, γιατί πήγε εκεί, ε, για την ιδεολογία, γιατί ήθελε να... Τον ήλκε γενικά τον τζιχάντα, ας πούμε. Ε, δεν τον βοήθησε καμία ομάδα. Ε, μόνος του πήγε. με τα χρήματα που είχε πέρασε από κάτω από όλα τα ραντάρα που, που θα μπορούσαν να το ψάχνουν. Για την Europol, ε, την ενεργητική προσπάθεια που θα πρέπει να κάνει η Europol. Τα κράτη-μέλη δεν θέλουν η, κράτη, η Europol να κάνει δράσεις, οποιασδήποτε δράση σε αυτό το τομέα. Η πρότασή μου ήταν να υπάρξουν εμπειρογνώμονες στην εποπτεία και παρακολούθηση του ίντερνετ, των παράνομων αυτών ε, ιστοσελίδων του τζιχάντ και των την εποπτεία επίση των κοινωνικών ε, δικτύων. Με αυτόν τον τρόπο θα κάνουμε και οικονομίε κλίμακα. παρά να κάνουν όλα τα κράτη-μέλη, το καθένα, α πούμε, έλεγχο του ίντερνετ. Τώρα, για την ερώτηση της ε, Σάρα Λάτφορντ, για το PNR και το profiling. Κατάλαβατε πολύ καλά τι είπα για τη χρήση του PNR, για την ε, δυνατότητα που μας δίνει να καταλάβουμε πού πρέπει να ξεκινήσουμε την επόμενη, το επόμενο screening. Ε, ούτως ή άλλως ε, οι αρμόδιες υπηρεσίες αυτή τη δουλειά έχουν, να ψάξουν οτιδήποτε είναι ύποπτο. Η δεύτερη, ο δεύτερος έλεγχος μπορεί να οδηγήσει κάλλιστα σε τίποτα. Τότε αυτές οι πληροφορίες, αν δεν οδηγήσουν σε τίποτα, σβήνονται. Αλλά όταν υπάρχει υπο, υποψία αμέσως μετά την ε, συλλογή των δεδομένων μπορεί να αρχίσει να σημαίνει το καμπανάκι. Αυτό είναι το θέμα. Θα αρχίσει να σημαίνει αμέσως ή πιο αργά θα αρχίσει να σημαίνει. Και αυτό είναι θέμα συναπόφασης ε, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για την πρόληψη. Κύριε Χιμένες, χαίρομαι που η κυρία Μάλστρομ ασχολείται με την Μάλστρομ ε, προσπαθεί να δημιουργήσει αυτό το δίκτυο για την ε, συνειδητοποίηση κατά της ριζοσπαστικοποίηση. Εγώ συμμετέχω σε πολλέ συνεδριάσει σε διεθνέ επίπεδο για τέτοια θέματα. Κανένα δεν, έχει βρει, δεν βρήκε την πανάκια. Μόνο με, τις, με το να δούμε ποιε είναι οι καλέ πρακτικέ, με τη δικτύωση των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, δεν μιλάω καν για βέλτιστε πρακτικέ, έτσι. Είναι υπερβολικό να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο να δούμε τι λειτουργεί, εν πάση περιπτώσει, απλώ. Αυτή είναι μια καλή απόφαση. Τον Νόβι θα γίνει και μια υπουργική διάσκεψη φέτο. Θα προσπαθήσουμε να ανταλλάξουμε αυτέ τι καλέ πρακτικέ. Η Αλκάιδα τώρα. Ε, όσο μειώνεται, θα μειώνεται και ο αριθμό των ε, επιθέσεων. Νομίζω συνολικά ναι. Αλλά φοβάμαι ότι άλλοι θα τη μιμηθούν. Φυσικά, ε, με βάση τα όπλα που υπάρχουν, μπορούμε να φτιάξουμε εκρηκτικά. Και ξέρετε ότι με τον πόλεμο των Βαλκανίων, ας πούμε, φτάσαν πολλά τέτοια όπλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με το ίντερνετ μπορούν να εμπνευστούν διάφοροι έτσι απογοητευμένοι, θέλουν να κάνουν, ας πούμε, ό,τι κάνει προηγούμενοι. προηγούμενοι. Θέλουν να κάνουν όπως έκανε ο Μέρα, ας πούμε. Ε, φοβάμαι, ας πούμε, τον μιμητισμό και την, την έμπνευση που δημιουργούν. Για την ναι, ΕΤΑ. Δεν μπορώ να σας πω κάτι έξυπνο για την αξιοπιστία της κατάπαυσης του πυρός. Δεν είμαι εμπειρογνώμονας για την ΝΕΤΑ. Από ό,τι που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, συχνά ρώτησα τους Ισπανούς ε, και τις Ισπανικές αρχές αν πρέπει να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Προσπαθούν οι Ισπανοί να τα αντιμετωπίσουν μόνοι τους με τη Γαλλία και με την ε, Πορτογαλία. Έχουμε βεβαίω το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, Έχουμε διάφορα πράγματα για να διευκολύνουμε τη συνεργασία. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν για την καταπολέμηση της ΕΤΑ. Ο νέος Υπουργό ε, στην πρώτη του αρμόδιος Γάλλος Υπουργό, έκανε έκκληση για διάλυση της ΕΤΑ και για παράδοση των όπλων. Η ΕΤΑ εξακολουθεί όμως να υπάρχει. Οι γαλλικές αρχές ε, είναι αποφασισμένε πάντω να βοηθήσουν την ε, ισπανική κυβέρνηση για να διαλύσει την ΕΤΑ. Ούτως ή άλλως αυτή η συνεργασία έχει δώσει και καλά αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Αυτά. Σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά, κυρία Δεκερκό για τις αφέστατες απαντήσεις. Πριν τελειώσουμε, βλέπω ένα χέρι υψωμένο. Τι θέλεις, τι θέλετε κυρία Φλότχο, ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ε, με καταλάβατε για την υπόθεση μέρα. Βασικά γι' αυτό ήρθατε. Παρότι εντάξει, θίξαμε και πολλά άλλα θέματα και σωστά και καλά κάναμε. Εγώ σας έλεγα ότι όχι ότι μας διέφυγε, διέλαθε της προσοχής μας ο Μέρα, αντίθετα, τον είχαμε στην προσοχή μας. Και το γεγονός ότι πήγε στο Ισραήλ με τη βοήθεια των μυστικών υπηρεσιών, ότι πήγε σε στρατόπεδο τη εκπαίδευση και έφερε πληροφορίε, όλα αυτά τα ξέραμε. Δεν ισχύουν αυτά που μας ε, λέτε. Και σε καμία περίπτωση η υπόθεση μέρα δεν χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσουμε, ας πούμε, το φαινόμενο της ε, ριζοσπαστικοποίησης. Μην χρησιμοποιείτε αυτή την υπόθεση που είναι αμφίσιμη απόλυτα. Την ξέραμε αυτή την ιστορία. Αυτό ήταν και το πρόβλημα, ότι το ξέραμε και όμως συνέβη ότι συνέβη. Εσείς αναφέρατε τη Frontex. Τι δουλειά έχει η Frontex αυτήν την ιστορία. Όπως είπατε κι εσείς, έφυγε με θεώρηση, με πληρωμένα εισιτήρια. Τι δουλειά έχει η Frontex εκεί μέσα. Πώς μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Δεν σας καταλαβαίνω. Νομίζω ότι τα ανακατεύετε όλα. Είναι γκροτέσκο αυτό που κάνετε. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω έτσι. Άλλο σχόλιο κύριε Κέρκοφ. Κοιτάξτε, αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι Δεν είναι όλοι ε, οι τζιχαντιστές τρομοκράτες μερά. Δεν είναι ίδιοι όλοι με το μερά. Εσείς θέλατε να σας ε, εκφέρω μία κρίση. Δεν είναι ο δικός μου ρόλος για την υπόθεση μεράχνια να σας πω αν ε, ήταν σωστή ή όχι η δράση των υπηρεσιών. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μου. Ο ρόλος μου είναι να δω τις διαφορές ε, στις διάφορες επιθέσεις, ποιες απετράψαν, ποιες ε, απετεύχθησαν, ε, να κάνω κάποιες σκέψεις, να κάνω κάποιες συγκρίσεις και κάποιες προτάσεις για κάποιες πολιτικές εξελίξεις. Και η ίδια η γαλλική κοινωνία θα κρίνει, πιστεύω, στην προκειμένη περίπτωση, εάν όπως είπατε ήταν πράγματι όχι πληροφοριοδότης της των γαλλικών μυστικών υπηρεσιών εγώ τα διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά, αλλά δεν μπορώ, ούτε και είναι ο ρόλος μου να κάνω έρευνα πάνω σε αυτό και δεν μπορώ να σας κάνω και μια ευφύ κρίση. Υπάρχουν οι λεγόμενοι clean skin. Δεν μου αρέσει καθόλου ε, αυτός ο όρος, αλλά έτσι λένε οι Αμερικάνοι. Είναι άνθρωποι οποίοι είναι υπεράνω πάθησης υποψίας, ας πούμε, και ε, γι' αυτό και δεν τους καταλαβαίνει κανένας. Ε, δεν μπορεί να εντοπίσει τη δράση τους. Δεν θέλω να κάνω καμία παρατήρηση, γιατί είναι προφανές για ποιο λόγο, επάνω στο πώς δρούν οι γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Απλά είπα ότι υπάρχουν κάποια θέματα που πρέπει να... Κάποια ερωτηματικά το πρέπει να απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Να ευχαριστήσω μια ακόμη φορά τον κύριο Ντεκερκόφ. Θα συνεχιστεί σίγουρα η συζήτηση και η δράση μας ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Όπως σας είπα λοιπόν και πριν, όταν ξεκινήσαμε, σε ΣΤΟΠΑ, στην αίθουσα θέλω να παραμείνουν όσοι μπορούν να παραμείνουν για τις συνεδρίες των συντονιστών. Όσοι δεν δικαιούνται να παραμείνουν, να αποχωρήσουν παρακαλώ. Σε πέντε λεπτά θα ξεκινήσει η συνεδρία των συντονιστών. Θα δώσουμε έτσι δύο-τρία λεπτά στους συντονιστές για να τακτοποιηθούν, ε, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά λοιπόν μετά σε πέντε λεπτά.